Eh, Συνάδελφοι, σας παρακαλώ πολύ, ας ε, αρχίσουμε με τις εργασίες μας. Παρακαλώ καθίστε έτσι ώστε να μην καθυστερούμε με την έναρξη των εργασιών μας. Όπως ε, γνωρίζετε, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης έχει κάπως αλλάξει σε σχέση με την ε, αποστολή των εγγράφων την προηγούμενη εβδομάδα και προβλέπεται ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη η ανταλλαγή απόψεων με τον Πίτερ Φάιτ, τον ε, ειδικό εκπρόσωπο για θέματα του πεδίου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι θα μας ενημερώσει σήμερα για την κατάσταση σε αυτή την ευπαθή ζώνη των Βαλκανίων. Θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στον δόκτορα Φάιτ να σας ε, μιλήσω για το πρόγραμμα αυτών των ημερών και ιδιαίτερα για την αυριανή μας συνεδρίαση. Όπως γνωρίζετε, αύριο το πρωί έχουμε την ψηφοφορία για το σχέδιο σύστασης ως προς την εταιρική σχέση και συνεργασία με το Τατζικιστάν και τον προπολογισμό του 2010. Αύριο το απόγευμα θα γίνουν οι ψηφοφορίες και θα πρέπει να το θυμόσαστε και να να φέρετε και την ηλεκτρονική σας κάρτα αύριο το απόγευμα στις 3 για τις ψηφοφορίες, την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ήθελα να πω ότι αύριο θα γίνει και η διάσκεψη του Διευρυμένου Προεδρίου μετά τις εργασίες της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι κατά την συνεδρίαση αυτή υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες εκτός από τα δανέζικα και τα μαλτέζικα. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη διερμηνία και από αυτές τις γλώσσες. Μία άλλη ανακοίνωση τώρα. παράλληλα με τη συνεδρίαση αυτή, στα πλαίσια της ΔΕΒΕ διενεργείται ακρόαση για τον διορισμό του Επιτρόπου μετά τον Λουί Μισελ, τον κύριο Κάρνβον Κούκτ. Η ΑΦΕΤ εκπροσωπείται στην ακρόαση αυτή δια του Φιωρέλο Προβέρα, πρώτου Αντιπροέδρου και από την κυρία Χάουταλα ε, που εκπροσωπεί και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 5η ε, στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι θα έχω μία συνάντηση με τον ε, ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ΚΕΠΑ, Χαβιέ Σολάνα, και βεβαίως θα σας ε, ε, θα μιλήσω για αυτή τη συνάντηση στην επόμενη συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρείου. Επίσης, τη Δευτέρα στις 7 του μηνός θα συμμετάσχω στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργανώνει η Σουηδική Προεδρία υπό τον ε, Υπουργό Μπίλτ στο Γκέτλαντ και στην ημερήσια διάταξη υπάρχει και η ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα, τα διατλαντικά θέματα, το Αφγανιστάν και η ειρηνευτική επίλυση του Μεσανατολικού. Θα ήθελα να κάνω μία ε, εισήγηση ως προς την παρέμβαση του Πίτερ Φάιτ, ο οποίος είναι ειδικό αντιπρόσωπος για θέματα κοσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη μας χαρά σας έχουμε για άλλη μια φορά μαζί μας. Ήδη μας είχατε μιλήσει κατά την προηγούμενη θητεία και η παρουσία σας όπως ορίστηκε για την αναθεώρηση των προγραμμάτων μας, ε, γίνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική στιγμή διότι ε, γνωρίζετε ότι προετοιμάζονται οι δημοτικές εκλογές στο Κωσυφοπέδιο για τις 15 Νοεμβρίου, άρα ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για τη γνώμη σας ως προς την προπαρασκευαστική διαδικασία αυτής της εκλογικής αναμέτρησης. Ελπίζουμε να συνεισφέρουμε και εμείς όπου χρειαστεί και ελπίζουμε να διενεργηθούν οι εκλογές με επιτυχία. Όπως γνωρίζετε, δόκτωρα Φάιτ, το Κοινοβούλιο είχε εκφραστεί δύο φορές για την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου υπό την αιγίδα του Μάρτι Αχτισάρη. Επειδή οι επόμενες εκλογές είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή ε, υπάρχει άμεση επαφή με τον πολίτη, έχει σημασία να δούμε πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα εξελιχθεί αυτό το αμάλγαμα μεταξύ σερβικού πληθυσμού και άλλων πληθυσμών επιτόπου. Μιλάμε για ένα πολυεθνοτικό σύστημα, το οποίο είναι πολυσχηδές και ευαίσθητο και ελπίζουμε να μπορέσει να ενταχθεί πολύ σωστά σε αυτή την οριοθέτηση που έχει γίνει, δηλαδή μέσα στα πλαίσια το, του, άμεσου συσχετισμού μεταξύ τοπικών αρχών και πληθυσμού. Βεβαίως γνωρίζετε ότι η EULEX είχε διαδραματίσει πολύ μεγάλο ρόλο στο κοσυφοπέδιο. Βρίσκεται σε λειτουργική φάση αλλά σε ορισμένους θυλάκους ε, στο βόρειο τμήμα της χώρας ήταν δύσκολο να αναλάβουμε αυτό τον αποφασιστική σημασίας ρόλο. Βεβαίως θα έχουμε και αμεσότερες πληροφορίες και γνωρίζω ότι έγιναν άμεσες επιθέσεις σε ευρωπαϊκά οχήματα. Θα ήθελα να μας πείτε πώς έχει το ζήτημα. Μακρηγόρησα όμως σε σχέση με θέματα τα οποία θα μας αναπτύξει ο Δόκτωρ Φάιτ και αφού τον ευχαριστήσω άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά θα ήθελα να του δώσω το λόγο. Grazie, signor presidente. Ευχαριστώ πολύ για τα ευγενή λόγια τα οποία μου απευθύνατε και θα ήθελα να διαβεβαιώσω τα μέλη της Επιτροπής και εσάς ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ ενώπιον του νέου Κοινοβουλίου και της νέας Επιτροπής. Την τελευταία φορά ήρθα το Φεβρουάριο και θα βασιστώ στις εκτιμήσεις μου, στις αξιολογήσεις μου για να σας παρουσιάσω την κατάσταση έτσι ως έχει στο κοσυφοπέδιο. Έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις εξελίξεις στο κοσυφοπέδιο και θα σας μιλήσω για την πρόοδο η οποία έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών αλλά και για τα προβλήματα τα οποία, στα οποία έχουμε προσκρούσει στο δρόμο μας. Το κοσυφοπέδιο έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις για τους επόμενους μήνες και θα προσπαθήσω να αξιολογήσω τις προκλήσεις αυτές εδώ σήμερα. Θα εστιαστώ κυρίως στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοσυφοπέδιο και θα σας πω μερικές σκέψεις για τις δικές μου προσπάθειες να συντονίσω και να προωθήσω τους στόχους της Ένωσης στην εκτέλεση της εντολής μου, είμαι ειδικό αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνω πολλή προσπάθεια για να αντικατοπτρίζω τις θέσεις όλων των κρατών μελών σε σχέση με το Κωσυφοπαίδιο. Κύριε Πρόεδρε, πολύ συχνά η προσοχή μας επισύρεται από τις ε, καθημερινές ε, ασχολίες. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για τις γενικές εξελίξεις στο κοσυφοπαίδιο. Εάν ε, δούμε την εποχή όταν πρωτοδιορίστηκα ειδικό αντιπρόσωπος τον Φεβρουάριο 2008, θα πρέπει να προσπαθήσω να κάνω μια σύγκριση με το σημερινό κοσυφοπέδιο. Έχουμε εδώ υγιή βελτίωση σε πάρα πολλούς τομείς και παρά ε, την εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται με συνεχείς προσπάθειες των αρχών να βελτιώσουν ε, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των πολιτών. Τους πρόσφατους μήνες το Κωσυφοπαίδιο έχει ε, κάνει ορισμένα σημαντικά επιτεύγματα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει τώρα ιδρυθεί και εγγενιαστεί. Το Κωσυφοπαίδιο κλήθηκε να γίνει μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας και οι αρχές έχουν προχωρήσει με βήματα ούτω ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα κριτήρια της ευρωπαϊκά διακυβέρνησης και ταυτόχρονα να να έχουν μέτρα αυτονομίας και ευκαιρίες για διάφορους να ενταχθούν στην πολυεθνική κοινωνία. Για να συμπληρώσω αυτή την εικόνα, το κοσυφοπέδιο και η καθημερινή ζωή του λαού με μερικές εξαιρέσεις έχουν ε, παραμείνει άφικτες από την βία και την ένταση την μεταξύ των εθνοτήτων. Στο Βόρειο-Ατλαντικό Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι η αποστολή και η ΦΟΡ θα έπρεπε να μειώσει την παρουσία της και νομίζω ότι αυτό αντανακλά την αξιολόγηση της διεθνούς κοινότητας ότι το περιβάλλον ασφαλείας στο Κωσυφοπαίδιο και στην περιοχή βαθμιαία αποκτά υψηλή σταθερότητα. Όντως υπάρχουν ορατά παραδείγματα αυτής της τάσης και θα ήθελα να αναφέρω μόνο μερικά από αυτά. Στην Πρίστινα η σερβική γλώσσα ομιλείται στους δρόμους και αυτό είναι καθημερινό συμβάν. Στο Δήμο του Καρμενίτσα έχουμε αγορές όπου οι Σέρβοι και οι Αλβανοί πουλούν τα προϊόντα τους ο κοντά δε. Και τέλος μια ομάδα πολιτικών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης των κοινοτήτων των Σερβικών και Αλβανικών στη Μητροβίτσα έχουν ετοιμάσει ένα φόρουμ για ε, να έχουν μια διάσκεψη μιας διηρημένης πόλης του χρόνου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η συμφιλίωση έχει επιτευχθεί ότι η διαδικασία δεν χρειάζεται συνεχή βοήθεια από το εξωτερικό. Οι διαφορές ανάμεσα και εντός των κοινοτήτων παραμένουν, αλλά οι διαφορές αυτές μειώνονται βαθμιαία με διαδικασίες δημοκρατικές και με θεσμούς δημοκρατικούς. Επειδή το κοσυφοπέδιο συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν περίπου όλα τα σκέλη των διαφόρων λειτουργιών πολιτικών και διοικητικών υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ούτω ώστε να πραγματοποιηθεί πραγματική πρόοδο για να υπάρξει πραγματική κοινοβουλευτική ε, διακυβέρνηση, καλή διακυβέρνηση. Το κοσυφοπέδιο έχει τώρα τους βασικούς θεσμούς με ευθύνες να προστατεύσουν τα δικαιώματα των λαών κόμμα, όπως είπα και το Συνταγματικό Δικαστήριο, το γραφείο του συνηγόρου του πολίτη και το, το δικαστικό συμβούλιο, για να σας αναφέρω μόνο μερικούς από αυτούς τους θεσμούς. Ωστόσο, τα όργανα αυτά θα πρέπει να ε, ενισχυθούν και να εκπληρώνουν ε, το έργο τους ε, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του κοσυφοπεδίου. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών στον τομέα αυτό θα είναι προς του λαού του Κωσυφοπεδίου, ε, κυρίως ε, για τις ε, επιθυμητές βελτιώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων και συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα ήδη το Φεβρουάριο, έχω την πρόθεση να ενθαρρύνω ανανεωμένες προσπάθειες ούτω ώστε ο ρόλος του Κωσυφοπεδίου να προωθηθεί διεθνώς για να βελτιωθεί η ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα αυτή. Η συνέλευση έχει δεσμευθεί για τις μεταρρυθμίσεις, τις θεσμικές, ε, οι οποίες συνεχίζονται στο κοσυφοπέδιο. Ωστόσο, θα πρέπει ε, να επιτύχει τον πλήρη ρόλο τον πολιτικό του κοσυφοπεδίου. Η συνέλευση πρέπει να προωθήσει την συμμετοχή της στην λήψη αποφάσεων και να βελτιώσει το επιπτικό έργο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί λογοδοσία και διαφάνεια. Θα ήθελα να καλέσω αυτήν τη διακεκριμένη επιτροπή, την αξιότιμη επιτροπή, να υποστηρίξει αυτή τη ε, διαδικασία, να, ούτως ώστε να περιληφθούν πλήρως οι μειονότητες στην πολιτική ζωή, διότι αυτό απαιτεί ε, σημαντικές προσπάθειες αφοσίωση από πλευράς ε, των αρχών του κοσυφοπεδίου σε συνεργασία με τη διεθνή κοινωνία και βεβαίως με την κοινωνία των πολιτών στο ίδιο το Κωσυφοπέδιο που θα είναι απαραίτητος εταίρος ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτή η συμπερίληψη όλων στην πολιτική διαδικασία. Το Φεβρουάριο, κύριε Πρόεδρε, ανέφερα ότι η σταθερότητα είναι στρατηγικός στόχος που πρέπει να επιδιεχθεί ε, σε συνεργασία με τις αρχές του Κωσυφοπεδίου. Πάντοτε η αρμονία δεν είναι τέλεια. Αυτή η εταιρική σχέση έχει, έχει γίνει μια στερεά συνεργασία όπου οι αρχές του Κωσυφοπεδίου έχουν επενδύσει πάρα πολλές προσπάθειες και δέσμευση αν οι δημοκρατικές διαδικασίες ήσουν να παρέχουν πολιτική σταθερότητα και μηχανισμούς για την διευθέτηση των διαφορών στο κοσυφοπέδιο, νομίζω ότι τότε ο κίνδυνος έντασης θα εξακολουθήσει να μειώνεται όλο και περισσότερο, να φθήνει. Ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι ε, με απασχολούν πολλά πράγματα. Με απασχολεί ε, η, ε, η κατάσταση των πολιτικών ηγετών ε, και ε, για το πώς ε, το κοινό δέχεται την διεθνή παρουσία στο Κωσυφοπέδιο ακόμα και αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οδηγεί σε βανδαλισμούς, σε βία, σε μια κακή ατμόσφαιρα που είδαμε κάποιες μέρες. Τούτων λεχθέντων, κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο κύριος εταίρος για το λαό του Κωσυφοπεδίου με την διακήρυξη της πλήρους ικανότητας της αποστολής Γιούλεξ, η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναβαθμιστεί. Η αποστολή Γιούλεξ τώρα εποπτεύει και συμβουλεύει την αστυνομία του Κωσυφοπεδίου σε όλους τους τομείς του κράτους δικαίου. Η πρόοδος μέχρι τώρα είναι ικανοποιητική στον τομέα αυτόν αλλά το κοσυφοπέδιο έχει ακόμα μεγάλο δρόμο μπροστά του και οι αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν να μπορεί η Γιούλεξ να συνεχίσει την αποστολή της με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Οι προσπάθειες μείωσης του οργανωμένου εγκλήματος είναι μεγάλη πρόκληση για τις αρχές του κοσυφοπεδίου. Αυτό θα απαιτήσει και πάλι την πλήρη υποστήριξη των αρχών και βεβαίως των τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εστιάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Το οργανωμένο έγκλημα δεν σταματάει στα σύνορα. Η πραγματική πρόοδος στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να συνεχιστεί να προωθηθεί βάση μιας περιφερειακής προσέγγισης. Οι προκλήσεις της Ιούλεξ στον τομέα του κράτους δικαίου είναι πολύ περίπλοκες στο βόρειο μέρος του ποταμού Ήμπαρ. Η Γιούλεξ έχει κάνει ε, βήματα προόδου με, την, ε, με ορισμένες τελωνιακές δραστηριότητες ε, στην πύλη 1 και 31 στο βορρά. Αυτό θα αρχίσει, αυτές οι προσπάθειες θα αρχίσουν να αποφέρουν καρπούς και θα αυξηθούν με την ενισχυμένη παρουσία τις επόμενες εβδομάδες. Παρ' αυτά, θα χρειαστούν σοβαρές προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στο Βορρά και να εξασφαλιστεί η καλή εκτέλεση, ε, πραγμάτωση του κράτους δικαίου. Ενώ η Ιούλεξ θα ενισχύει τις δραστηριότητες της στο Βορρά, είμαι ε, πεπισμένος ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνεται όλο και πιο αισθητά αναγκαία για να υποστηρίξει την αποστολή της Γιούλεξ. Το κοσυφοπέδιο ετοιμάζεται για τις πρώτες εκλογές που θα ακολουθήσουν μετά την μονομερή ε, διακήρυξη ανεξαρτησίας στις 18 Φεβρουαρίου 2008. Ο Φάτμιε Σέντιου, ο πρόεδρος, ανήγγειλε ότι τοπικές εκλογές, δημοτικές εκλογές ε, για δήμους ε, και συνελεύσεις ε, δημοτικές θα λάβουν χώρα στις 5 Νοεμβρίου φέτος. Ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή Εκλογική του Κωσυφοπεδίου να κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες ούτως ώστε να γίνουν αυτές οι δημοτικές εκλογές στο Κωσυφοπαίδιο. Εφόσον τα μέσα τα τοπικά αυτής της Επιτροπής είναι ακόμα περιορισμένα, χρειάζεται τεχνική υποστήριξη από διεθνείς πρωταγωνιστές, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Κωσυφοπέδιο θα υποστηρίξει και θα εκπαιδεύσει την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή για να προετοιμαστεί για τις εκλογές του 2009, ενώ έχουμε και βοήθεια Ηνωμένων Πολιτειών για πρόσθετες δραστηριότητες. Η Επιτροπή αυτή εκλογική ε, ζήτησε ορισμένες οργανώσεις περιφερειακές και ευρωπαϊκές να παρακολουθήσουν ε, τις εκλογές, να είναι παρατηρητές. Ελπίζω αυτό να γίνει, διότι, διότι μια μια διαδικασία δημοκρατική και διαφανής εκλογική είναι πρωταρχική σημασίας για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη του κοσυφοπεδίου ως σύγχρονη κοινωνία δημοκρατική και πολυεθνική. Οι δημοτικές εκλογές είναι σημαντικές για την τοπική αντιπροσώπευση και την παροχή υπηρεσιών σε όλες τις κοινότητες του Κωσυφοπεδίου. Οι διάφορες σχέσεις δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τα δικαιώματα των πολιτών να συμμετέχουν σε δημοκρατικές διαδικασίες και να εκπροσωπούνται δέοντος στο τοπικό επίπεδο, στο δημοτικό επίπεδο. Οι επόμενες εκλογές οργανώνονται σε μια εποχή όπου ε, γίνονται σημαντικές τοπικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις αποβλέπουν ε, στην συμπερίληψη και συμμετοχή όλων των κοινοτήτων στα θεσμικά όργανα του κοσυφοπεδίου, ούτως ώστε να υπάρξει ε, μια διαβίωση σταθερή και βιώσιμη για όλους. Ε, η Δήμη με πλειοψηφία ε, σερβική ε, έχουν εξελιχθεί και θα έχουν δικαιώματα αυτονομίας και θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των Σέρβων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η διαδικασία ε, για αυτές τους δήμους όπου θα υπάρχει ε, πλειονότητα Σέρβων είναι μέρος της διαδικασίας αποκέντρωσης του κοσυφοπεδίου. Αλλά βεβαίως Βασικά πρόκειται για μια προσπάθεια των αρχών του Κωσυφοπεδίου ε, να τίνουν χείρα βοηθείας στους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Βεβαίως η επιτυχία αυτής της προσπάθειας ενέχει τεράστια σημασία για το μέλλον του πολυεθνικού Κωσυφοπεδίου η αποκέντρωση θα επιτρέψει στο, ε, στο κοσυφοπέδιο μια συμφιλίωση με τις μειονότητες, μια ευρύτερη αντιπροσώπευση σε τοπικό επίπεδο της μειονότητας των Σέρβων θα επιτρέψει σε αυτήν την μεγάλη μειονότητα που ζει στο κοσυφοπέδιο να έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την διαχείριση των υποθέσεών της. Αυτό περιλαμβάνει θέματα τα οποία είναι κλειδιά για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, όπως η υγεία, η παιδεία, όπως επίσης η προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Ορθοδόξων Σέρβων ως ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία σε στενή συνεννόηση με τη διεθνή κοινότητα, οι αρχές του Κωσυφοπεδίου προσπαθούν να αξιολογήσουν πόσες από, πόσοι από αυτούς τους Δήμους θα είναι σε θέση να λάβουν μέρος στις εκλογές του Νοεμβρίου. Προφανώς σε αυτές τις εκλογές η συμμετοχή των πολιτών, το βαθμό συμμετοχής θα είναι ένα σημαντικό κριτήριο. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση της Σερβίας θα ενθαρρύνει τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Κύριε Πρόεδρε, οι προκλήσεις για το λαό του Κωσυφοπεδίου δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν χωρίς πρόοδο στην ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία, οικονομική και εμπορική συνεργασία. Σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και των δικαιωμάτων της κοινότητας των Ρωμά. Ε, προώθηση των μέτρων για την ένταξη στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα επιτρέψουν καλύτερη συνεργασία στην ευρύτερη ε, περιφέρεια με την υποστήριξη της ε, διεθνούς κοινότητας στον τομέα του κράτους δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτελεστεί πρόοδος ε, στην συνεργασία με τη Σερβία, στους τομείς της αστυνομίας και των τελωνίων, όπως τονίστηκε από τις, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ελευθεροποίηση των, του θέματος των θεωρήσεων. Το κοσυφοπέδιο έχει κάνει σημαντική πρόοδο για τους δημοκρατικούς θεσμούς και μηχανισμούς και για την βελτίωση της ζωής των πολιτών. Έχει αρχίσει το ταξίδι προς την εδραίωση αυτών των επιτευγμάτων με μεταρρυθμίσεις της τοπικής κοινωνίας, με έργα υποδομής και με βελτιώσεις στην οικονομική διακυβέρνηση. Έχει αρχίσει να οικοδομεί μια πραγματική εταιρική σχέση ε, με την Ευρωπαϊκή Αποστολή Κράτους Δικαίου. Θα έχουμε λοιπόν εδώ την πρώτη δοκιμασία, το πρώτο τεστ εκλογικό τον Νοέμβριο. Αυτό θα είναι επίσης μια ευκαιρία ε, για να δοκιμαστεί αυτή η αυτο, ε, αυτονομία, η αυτοδιάθεση που προσφέρεται στους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Έχουμε ακόμα σήμερα προκλήσεις, όπως είπα. Το κοσυφοπέδιο έχει ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσει προτού πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή του προοπτική. Θα χρειαστεί ισχυρή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις τα επόμενα χρόνια. Αλλά βάσει αυτής της έκθεσης και στενής συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου, ο λαός του Κωσυφοπεδίου θα μπορέσει να αισθανθεί ότι ε, θα έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το ταξίδι που έχει αρχίσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστούμε δόκτωρα Φάιτ για την ε, διεξοδική αυτή παρουσίαση και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν Εάν συμφωνείτε, επειδή προσπαθούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας για την ημερήσια διάταξη, θα ήταν σκόπο να έχουμε τρεις παρεμβάσεις και την απάντησή σας στη συνέχεια και μετά αν έχουμε λιγότερο χρόνο τότε θα συγκεντρώσουμε περισσότερες ερωτήσεις και εσείς, ε, δόκτωρα Φάιτ, θα μπορέσετε να μας απαντήσετε πιο συνοπτικά. Η κυρία Πακ ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον Πίτερ Φάιθ. Έλειπα όταν μιλήσατε για τις ε, εξελίξεις και τις πρόοδους, γιατί όταν ενημερωνόμαστε κυρίως για τα κακά μαθαίνουμε και χαίρομαι για τα καλά που απαριθμίσατε, που μας ενθαρρύνουν και μας ε, να δράσουμε υπέρ του κοσυφοπεδίου. Είπατε ότι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες, μιλήσατε για τη Μητροβίτσα. Πείτε μου, ποιος ελέγχει παρακαλώ τα σύνορα μεταξύ Κωσυφοπεδίου, Σερβίας, Μητροβίτσα, η Γιούλεξ μεταξύ, έχει λόγο ή άλλοι κάνουν, ε, ασκούν τον έλεγχο. Επίσης το σύστημα των θυλάκων ε, έχει αρθεί Δηλαδή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ακόμα οι θύλακοι αυτοί. πώς έχουμε προχωρήσει εδώ. Επίσης να μας πείτε και εσείς ως ειδικό απεσταλμένος πώς μπορείτε να ασκήσετε επιρροή ούτως ώστε η δουλειά επιτόπου, people to people, ε, μεταξύ τους να προωθήθει αυτό. Το έχουμε ε, πει, τουλάχιστον ε, γραπτός υπάρχει. Δηλαδή οι Σέρβοι και οι Αλβανοί θα πρέπει στις κοινότητες, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, να αρχίσουν να συνεργάζονται. Αυτό πρέπει να το προωθήσουμε επί τόπου. Τρίτον, βεβαίως θα θέλαμε να παρευρεθούμε και να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Πάντα το κάναμε και νομίζω ότι είναι υπέρ και των Αλβανών Κωσοβάρων και της μεγάλης πλειοψηφίας των, ε, των Σέρβων Κωσοβάρων να είμαστε εκεί και να αποδείξουμε εμπράκτος ότι θέλουμε να φροντίσουμε και εμείς και να συμβάλλουμε στο να αποβούν θετικές για όλους οι εκλογές. Επίσης, για το Βελιγράδι είπατε ότι ε, ενθαρρύνει τους Σέρβους. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Εγώ έχω ακούσει να τους αποτρέπει από τη συμμετοχή στις εκλογές. Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι προσπαθεί να κάνει κάτι και το Βελιγράδι προς αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να παίξουν το ρόλο τους και οι Σέρβοι και να μπορέσουν να πάρουν στα χέρια τους τη μοίρα τους στη χώρα στην οποία μένουν. Καλό θα ήταν αυτό. Τέλος, ε, ε, για αυτό που είπατε για το Κοινοβούλιο, και θέλω να καλέσω τα θεσμικά μας όργανα, ούτως ώστε οι συνάδελφοι από το Εθνικό Κοινοβούλιο να έρθουν εδώ και να δουλέψουμε μαζί πάνω σε επίκαιρα προβλήματα, ούτως ώστε να δουν πώς προχωράει η κοινοβουλευτική δουλειά και έτσι θα μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα και με την κυβέρνηση. Καλό θα ήταν αυτό να γίνεται και με την Κομισιόν. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία και στο μέλλον και παρακαλώ και ο Πρόεδρος να πάρει στα σοβαρά την έκκληση αυτή να στείλουμε μια επιτροπή παρακολούθησης των εκλογών εκεί. Ευχαριστώ. Λαμβάνω υπόψη την ε, παρατήρησή σας και θα την επαναλάβω στο τέλος της συζήτησης. Ο κύριος Βόποντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φάιθ για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ ρεαλιστικά νομίζω αυτά που μας είπατε και θέλω μόνο ένα πράγμα να υπογραμμίσω που αφορά τις εκλογές της 15 Νοεμβρίου γιατί όπως είπατε και εσείς είναι κέριο το ζήτημα. Αν υπάρξει πρόοδος, αν υπάρξει επιτυχία, θα σημειωθεί πρόοδος σε όλο το φάσμα στο κοσυφοπέδιο. Και προσυπογράφω αυτά που είπε η Ντόρις, αλλά ακόμα πιο θετικά για να το πω, πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τις επόμενες εβδομάδες να αξιοποιήσουμε τις επαφές μας. Ίσως μπορείτε να μας βοηθήσετε, εμείς δηλαδή ως Κοινοβούλιο και εσείς, να είμαστε σε μια μόνιμη επαφή αυτό το διάστημα, και με τους Σέρβους, τους Κωσοβάρους και τη Σερβική κυβέρνηση προφανώς, ούτως ώστε τουλάχιστον να ε, υπάρξει μια Σερβία και Σέρβοι που θα δεχτούν τις τοπικές ε, εκλογές ως προς τη σημασία τους για τις συνθήκες διαβίωσης της σερβικής μειονότητα ή του σερβικού πληθυσμού ή όπως και να το πούμε στο Πέδιο. Η ομάδα μας προφανώς στη διάσκεψη των Προέδρων θα στηρίξει το αίτημα και ο πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι και εκείνος θα το υποστηρίξει, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της 15ης, είναι θέμα των εβδομάδων που θα προηγηθούν, ούτως ώστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν εμείς ε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Δηλαδή, πέρα από την, ε, το νομικό ζήτημα, είναι στη Χάγη, αλλά πέρα από το νομικό ζήτημα, καλό είναι να επικεντρωθούμε στις συνθήκες διαβίωσης και στη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. Δεν, δεν είναι μόνο οι Αλβανοί και οι Σέρβοι, είναι και άλλοι. Και τα παραδείγματα που μας δώσατε πρέπει να κοινοποιηθούν παρακαλώ πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταδειχθεί ότι υπάρχουν αγορές, υπάρχουν χωριά όπου είναι δυνατή η συμβίωση και νομίζω ότι αυτή η Επιτροπή πρέπει να αξιοποιήσει τις επόμενες εβδομάδες πολύ αποτελεσματικά για να πείσει και να συμβάλλει στην επιτυχία αυτών των εκλογών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Βότσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φίθ για αυτά που μας είπατε σήμερα. Με ενδιαφέρον να άκουσα αυτά που είπατε για το φόρουμ της Μητροβίτσα και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για άλλου είδους πρόοδους επίσης στη Μητροβίτσα και το φόρουμ και σε ποιο βαθμό το φόρουμ αυτό ε, έχει απήχηση στους Σέρβους Κωσοβάρους. Επίσης η στάση του Βελιγραδίου απέναντί του ποια είναι από ό,τι βλέπετε. Υπήρξαν προσπάθειες ενδεχομένως να υπονομευθεί το έργο του φόρουμ. Επίσης, πείτε μας κάτι για τη στάση των κρατών μελών προς το έργο το δικό σας, ιδιαίτερα των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο και ποια κράτη-μέλη αν υπάρχουν βοήθησαν ιδιαίτερα πολύ ε, ε, προβλέποντας αποσπάσεις προσωπικού κλπ. Επειδή ο προϋπολογισμός σας από την Ένωση είναι τόσο μικρός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν για σας να σας βοηθήσουν αποσπασμένοι υπάλληλοι. Επίσης, ε, η αποστολή αυτή τι διάρκεια θα είναι, γιατί είχε προβλεφθεί η αποστολή σας μέχρι το 2010. Τώρα προφανώς θα πάρει σημαντικά περισσότερο χρόνο από αυτό. Εσείς πιστεύετε ότι θα ε, είστε ο εκπρόσωπος που θα τελειώσει το έργο ή θα σας διαδεχθεί κάποια στιγμή κάποιος άλλος. Ευχαριστούμε. Όπως συμφωνήσαμε, ο Δόκτωρ Φάιτ έχει το λόγο για να απαντήσει στις τρεις πρώτες ερωτήσεις και θα συνεχίσουμε με άλλες ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν, πρέπει να πω ότι με ενθαρρύνουν πάρα πολύ τα λεγόμενα της κυρίας Πακ και του κυρίου Σβόμποντα για τη σημασία των δημοτικών εκλογών. Και το ενδιαφέρον που καταδεικνύουμε όλοι για τις κοινότητες που θέλουμε να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος, ο στρατηγικός στόχος των αποστολών μου. Αυτό είναι και διευκρινίζω αμέσως τον κύριο Βότσον ότι αν και βρίσκομαι εδώ ως ειδικό ε, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστό ότι έχω και μια άλλη ένα, ε, ευθύνη. Όλα αυτά όμως ε, συμπλέουν αν θέλετε για να στηρίξουν το στρατηγικό στόχο που είναι η επίτευξη της ενσωμάτωσης των κοινοτήτων στο κοσυφοπαίδιο. Αυτό είναι θεμελιώδες προαπαιτούμενο για τη σταθερότητα στην οποία προσβλέπουμε στα Βαλκάνια, στη περιοχή και στο Κωσυφοπαίδιο. Ε, ένα συστατικό λοιπόν, ένα τακτικό πρώτο βήμα θα είναι να ενθαρρυνθούν οι Σέρβοι από εμάς να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αν και οι δύο διαδικασίες είναι χωριστές. οι δημοτικές εκλογές και η διαδικασία της αποκέντρωσης ε, εμπλέκονται και τρόπον να αλληλοεξαρτώνται γιατί θα πρέπει να Ε, με τις δημοτικές αρχές στους δήμους που θα μετασχηματιστούν και θα έχουν σερβική ε, πλειοψηφία. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να δει η σερβική πλευρά αυτή τη δυνατότητα, τόσο ώστε να γίνουν οι αποδέκτες των Δήμων με τα αυξημένα ε, δικαιώματα ε, αυτονομίας τους. Ενισχυμένα δικαιώματα. Ε, πρέπει να πω και χαίρομαι γι' αυτό ότι προχωρήσαμε σημαντικά με τη διαδικασία της αποκέντρωσης και ε, θεωρώ ότι με την καλή συνεργασία με τις αρχές, ε, δηλαδή το Υπουργείο Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στο Κωσυφοπαίδιο, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να ολοκληρώσουμε την ε, θέσμηση των ε, δημοτικών προπαρασκευαστικών ομάδων όπως λέγονται που αποτελούνται κυρίως από Σέρβους κοσοβάρους, ε, αξιωματούχους, ειδικού που θα προετοιμάσουν τους νέους δήμους ώστε να καταστούν αυτοί λειτουργικοί. Αυτό νομίζω θα το τελειώσουμε πριν από τις 15 Νοεμβρίου. Και είναι, θεωρώ, πολύ ισχυρό μήνυμα που αποστέλλεται προς τη σερβική κοινότητα αλλά και προς το Βελιγράδι, ότι δηλαδή οι εκλογές θα πρέπει να ε, θεωρηθούν μια θετική ευκαιρία που μπορεί να αξιοποιηθεί. Δεν είμαι σε θέση ε, να πω κάτι παραπάνω από εικασίες ε, σχετικά με το τι θέση θα πάρει το Βελιγράδι εν ώψη αυτών των νέων εξελίξεων. Επαναλαμβάνω όμως και πάλι ότι πολλά έχουν να κερδίσουν και αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομική θέση των μερών σε σχέση με το καθεστώς του Κωσόβου αν οι εκλογές αυτές επιτύχουν. Δηλαδή δεν θα επηρεαστεί το νομικό καθεστώς και το πώς αυτό πορεύεται. Ε, χαίρομαι που μπορώ να σημειώσω το, το ενδιαφέρον που εκφράσατε να συμμετάσχετε σε μια επιτροπή παρακολούθησης των εκλογών. Τώρα κάνω διαβουλεύσεις με την Κομισιόν σχετικά με το πώς θα οργανωθεί μια αποστολή παρακολούθησης, ε, τη απουσία του ΟΑΣΕ που είναι περιορισμένος ε, από την εντολή που έχει σε σχέση με αυτό. Πρέπει λοιπόν άλλος οργανισμός να αναλάβει και πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω άλλο θεσμικό όργανο από αυτό εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ο πλέον ενδεδειγμένος και κατάλληλος εταίρος στην εκλογική διαδικασία, δεδομένης της ευρωπαϊκής προοπτικής που έχει δοθεί στο Κωσυφοπαίδιο ως ε, τμήμα της περιοχής αυτής. Τώρα για τα άλλα συγκεκριμένα ερωτήματα, εδώ θα είμαι μάλλον συντομότερος. Η κατάσταση στο Βορρά ακόμα είναι πολύ σύνθετη. Η Ulex είναι στις δύο πύλες όπου γίνεται η καταγραφή των προϊόντων με την, υπό την εποπτεία της Ulex. Κατά τα άλλα, η κοσοβάρικη αστυνομία, ως επιτοπλίστων, η Σέρβια στη νομική, ε, παρακολουθούνται από τη Ulex και αντιμετωπίζουν κυρίως την πρόκληση της ανασυγκρότησης των κατοικιών στο Βίτακουτ και στο Κόρι σε αυτές τις δύο περιοχές που είναι κοντά στο βορρά της Μητροβίτσα. Ίσως ε, έχετε δει ε, κάλυψη από τα ΜΜΕ, υπάρχει όμως εδώ πρόβλημα βίας ε, πρέπει να αποκατασταθεί η σταθερότητα και οι δημοτικές εκλογές ελπίζομαι μεταξύ άλλων να βοηθήσουν να ε, ξεπεραστούν οι παράλληλες δομές και μετά δικαιώματα αυτονομίας που, που θα δοθούν στις κοινότητες, αυτές οι παράλληλες δομές σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταργούνται. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά, ιδιαίτερα εις ό,τι αφορά και τη βιωσιμότητα των θεσμών του κοσυφοπεδίου. Τώρα, για το φόρουμ, μπορώ μόνο να πω ότι τώρα έχουμε πολλαπλές επαφές με τους Σέρβους Κωσοβάρους, με την κοινότητά τους, αλλά και με μονομένα μέλη της, στη Μητροβίτσα. Και σύν το χρόνο ελπίζομαι και ίσως να έχει γίνει ήδη 10, να γίνει στις 15 Νοεμβρίου αρχή αλλά και μετά με, άμεσα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του Δήμου στο βορρά της Μητροβίτσα, όπως προβλέπει το οικιστικό πρόγραμμα, το συνεκτικό που έχει προταθεί από τους Σέρβους. Ο κύριος Βότσον με ρώτησε ε, για τη μελλοντική μου θητεία, αν θέλετε, και το ρόλο που θα παίξω στο Πέδιο στο μέλλον. Ε, αυτό πάντα είναι ένα επικίνδυνο ερώτημα. Ελπίζω ότι θα ε, μπορέσω ε, να ξανάρθω στη Σεβαστή Επιτροπή για να πω κι άλλο για το κοσυφοπαίδιο σχετικά με τις εξελίξεις, αλλά αυτά θα εξαρτηθούν η μελλοντική μου θέση θα εξαρτηθεί από την ε, ομόφωνη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών. Ε, γιατί εδώ υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποφασίστηκαν και συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του 2007, αρχές του 2008, δηλαδή υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης Κωσυφοπεδίου και ειδικότερα υποστήριξη της ενίσχυσης του κράτους δικαίου στο κοσυφοπέδιο και τα 27 κράτη-μέλη στήριξαν τις προσπάθειές μου και του, της, ε, τις ε, προσπάθειες του επικεφαλής της αποστολής Γιούλεξ του στρατηγού Ντεκερμαμπών και εγώ είμαι πολύ ευγνώμων σχετικά με τις προσπάθειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φάιντ. Τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο αρχίζοντας από τον κύριο Λούνατσεκ. Κύριε Λούνατσεκ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Λούνατσεκ. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω κύριε Φάιντ εξ ονόμας των Πρασίνων για την παρουσίασή σας και για ε, τη θετική πορεία του κοσυφοπηδίου και όχι μόνο τις δυσχέρειες που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν στη χώρα αυτή. Πολύ σωστά αναφερθήκατε στην ανάγκη να προωθήσουμε την οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στη χώρα, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν την αίσθηση ότι τους ανήκει η χώρα αυτή, μπορούν να εργαστούν εκεί και να παραμείνουν και δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα τους έτσι ώστε να έχουν καλύτερη τύχη, καλύτερη οικονομική τύχη σε άλλες χώρες. Εμείς στην Αυστρία, από όπου προέρχομαι, έχουμε πολλούς που προσέφυγαν σε μας και ακόμα προσπαθούν. Γι' αυτό παρακολουθώ την κατάσταση εκ του σύνεγγης. Κύριε Φάιτ, εξ ονόματος της ομάδας ε, υποστηρίζω αυτό που ήδη προελέχθη και που αναφέρατε και τώρα, δηλαδή να αποστείλουμε παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΑΣΕ θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι είναι ε, έκτακτη κατάσταση. Αυτό αφορά και τις ιδιαιτερότητες της χώρας. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή αποστολή. Η κυρία Πάκο, ο κύριος Φόμποτα και άλλοι το είπαν και ελπίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας και εσείς μιλήσατε για τις αστυνομικές αρχές και τη συνεργασία αυτή. Πόση ευρωπαϊκή βοήθεια χρειάζεται για την αστυνομία, διότι η αστυνομία ε, εξασφαλίζει την ασφάλεια, όταν βεβαίως είναι καλώς καταρτισμένοι. Εάν υπάρχει, αν υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις που δεν έχουν τη σωστή κατάρτιση, τότε οι πολίτες φοβούνται την αστυνομία. Μιλήσατε για το οργανωμένο έγκλημα επίσης και εδώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση ιδιαίτερα για τις γυναίκες στη χώρα. Ξέρουμε ότι η σωματεμπορία είναι κάτι που αφορά τις ε, γυναίκες και τα κορίτσια, κυρίως τις γυναίκες και τα κορίτσια και πολλές γυναίκες βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση γιατί δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση ούτε βεβαίως και εισόδημα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο λίγα περισσότερα στοιχεία για την ε, ενδεχόμενη πρόοδο σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να προσθέσω αυτό που ήδη είπε ο κύριος Φόμποτα. Άκουσα ότι το Βελιγράδι στέλνει προειδοποίησεις ε, τους, ως προς ε, του Κωσυφοπεδίου να μην συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές. Ελπίζω το Βελιγράδι να δει ότι οι δημοτικές εκλογές είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, είναι ένα ε, ένα μέτρο για να αναλάβουν τα πράγματα, να αναλάβουν δηλαδή ευθύνες. Αυτό αφορά του Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Τι προοπτικές βλέπετε σε σχέση με τη στάση του Βελιγραδίου έτσι ώστε να προτρέψει τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου να ψηφίσουν. Και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια τελευταία ερώτηση που ίσως είναι ευαίσθητη εσείς ε, είπατε ότι και μας είπατε ότι δεν είσαστε μόνο ε, ο Ευρωπαίος εκπρόσωπος και ξέρουμε το ICR, ICO, επειδή ε, είσαστε εκπρόσωπος του πολιτικού σκέλους και όχι του στρατιωτικού, προωθήθηκε μέσα σε αυτά τα πλαίσια η ανεξαρτησία του Κωσοφοπεδίου. Σε αυτή τη δυτή σας οντότητα βλέπετε να υπάρχει μια αντίφαση, δηλαδή από τη μία χρηματοδοτείται το ICR και από χώρε που δέχτηκαν την ανεξαρτησία όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς πρέπει να είσαστε ουδέτερος. Βλέπετε σύγκρουση συμφερόντων, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω, αλλά μου ελέγχθη ότι ίσως ε, ανακύψει πρόβλημα. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ, ο κύριος Βανόρτεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πίτερ Φέιθ που ήρθε σήμερα το απόγευμα και τον συγχαίρω κιόλα. Γιατί με μεγάλο επαγγελματισμό ανταπεξέρχεται στα καθήκοντα της δύσκολης αποστολής του. Το λέω αυτό πέρα από τις διαφορές μας σε σχέση με το καθεστώς του Κωσόβου. Η αποστολή Γιούλεξ είναι υπό την γίδα της ΕΠΑ ε, ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα και πολύ σημαντική δουλειά γίνεται και στα πλαίσια της πολιτικής υποστήριξης. Αλλά υπάρχουν κάποιες ε, σοβαρές αντιρρήσεις σε σχέση με τη στρατιωτική του ε, δραστηριοποίηση ή να μπαίνουν στρατιωτικές ταμπέλες σε πολιτικές αποστολές. Ανέφερες την K4 πολύ εμπαρόδο. Είναι περίπου 14.000 όμως ε, οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ στα πλαίσια της ΚΕΙΦΟΡ και περισσότεροι προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες γιατί το ΝΑΤΟ εν είναι ευρωπαϊκός οργανισμός πολλοί το ξεχνούν αυτό το πράγμα Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα πράγματα σε σχέση με το συντονισμό μεταξύ Γιούλεξ και ΝΑΤΟ γιατί λέτε ότι μειώνεται η αποστολή του ΝΑΤΟ. Αυτό τώρα τι προοπτικές έχει στο μέλλον, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Τώρα, σε σχέση με την αστυνομία του Κωσόβου, ε, έχετε συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό βέβαια ε, εισπράτεται με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή τους εκπαιδεύετε τους αστυνομικούς ή τους δίνετε συμβουλές γιατί, ε, πα, παρακολουθώντας τους τις αποστολές. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και μια εντολή εκπαιδευτική ως ε, τμήμα, αν θέλετε, των δραστηριοτήτων που πρέπει να κάνετε. Τι αστυνομία είναι αυτή. Είναι, ας πούμε, δύο διαφορετικές χωριστές, ξέχωρες αστυνομικές δυνάμεις ή είναι διακοινωτική αστυνομία στο Κόσοβο. Αναφερθήκατε και στη δικιά σας την εντολή. Η εντολή είναι για την αποστολή μέχρι το 2010. Ο Γκρέμ Βάτσον λέει δεν έχετε πολλά λεφτά. Νομίζω είναι 265 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα τα λεφτά. Για πόσο καιρό βλέπετε να χρειάζεται η αποστολή. Πόσο καιρό θα πρέπει να υπάρχει αυτή της κλίμακας η παρουσία στο κοσυφοπέδιο; Πιστεύετε δηλαδή ότι θα χρειαστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βανόρντεν. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Κύριος Χουντής, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, ενδιαφέρουσα η ενημέρωση για το κοσυφοπαίδιο. Όμως παραμένει ένα κεντρικό ερώτημα που ενισχύθηκε και από τα λεγόμενα του, του εισηγητή. Τελικά, η πολιτική, η βοήθεια, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά το στάτους του Κωσυφοπεδίου, προς τα που κατατείνει. Αφού πω για άλλη μια φορά ότι η θέση της ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς είναι κατά της ανεξαρτοποίησης του Κωσυφοπεδίου, έχουμε τη σημερινή εικόνα 62 χώρες κατά τα, την ενημέρωση που έχω να έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου, μεταξύ αυτών και ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα τίθεται, βλέπετε ότι μπορεί να ανακοπεί αυτή η πορεία ανεξαρτοποίησης που κατά την, ε, αναγνώριση της ανεξαρτοποίησης που κατά την άποψή μας εντείνει τις διαμάχες, δημιουργεί ένταση στην περιοχή, δημιουργεί κακό προηγούμενο αλλαγή συνόρων. Υπάρχουν δυνατότητες να υπάρξει μια νέα ειρηνευτική διαδικασία ούτως ώστε να βρεθεί μια λύση σύμφωνα με το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας που κατά την άποψή μας μπορεί να δώσει μια λύση που θα εξασφαλίζει τη σταθερότητα και στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Τι θα γίνει με το πρόβλημα των προσφύγων πολέμου που έφυγαν και τις δυνατότητες να επανέλθουν στις πατρίδες τους, στις αιστείες τους. Και το τελευταίο, ε, αναφέρθηκε, αναφέρθηκαν ορισμένα σημεία πόσο μας ανησυχεί το γεγονός ότι το Κωσυφοπαίδιο παραμένει χώρος οργανωμένου εγκλήματος με διακίνηση ναρκωτικών, σωματεμπορίας και τι μπορεί να γίνει σε αυτή την κατάσταση που αποτελεί, αν αληθεύουν οι πληροφορίες και αν έτσι είναι τα πράγματα, πληγή και για την ευρύτερη περιοχή και για την περιοχή της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χουντή. Θα ήθελα να δώσω για άλλη μια φορά το λόγο στον δόκτωρα Φάιτ για, μια, για την απάντηση στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Και μετά θα ομαδοποιήσω τέσσερις ερωτήσεις για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. νομίζω ότι εισαγωγικά πρέπει να διευκρινίσω και στην κυρία Λούνατσε και στον κύριο Μανόρντεν, κυρίως τον τελευταίο, ότι δεν είμαι επικεφαλής της, ε, της αποστολής Γιούλεξ για το κράτος δικαίου. Είμαι ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν δίνω εγώ τις εντολές, ε, απλώς ε, είναι πολιτικός συμβουλευτικός ρόλος μου, καθοδηγητικός πολιτικός. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση αν δεν θα μπορέσω να μπω στο βάθος των επιχειρησιακών ζήτηματων, ελπίζοντας ότι ο κύριος Ντεκερμαμπόν που είναι ο επικεφαλής της αποστολής Γιούλεξ, θα απαντήσει σε λεπτομερέστερες ε, ερωτήσεις. Ιδιαίτερα κυρία Λούνατσεκ. δεν έχω στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή μου σχετικά με την πρόοδο στην καταπολέμηση τη σωματεμπορία γυναικών, τη εμπορία γυναικών. Σε αυτό το στάδιο νομίζω ότι μπορώ να πω ότι επιτελείται πρόοδο, αλλά ακόμη δεν έχει εκριζωθεί το πρόβλημα και το κοσυφοπέδιο παραμένει χώρα διέλευσης ε, σε, από πολλές απόψεις, όχι μόνο για τα ναρκωτικά, αλλά και στην σωματεμπορία. Αυτό που θα έπρεπε να πω ίσως είναι ότι οι ε, αρχές ε, του κοσυφοπεδίου έχουν κάποια ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού φύλου. Να δώσω κάποια παραδείγματα. Ε, υπάρχει ε, μια ποσόστοση 30% για τις γυναίκες που επιθυμούν να ε, συμμετάσχουν στην συνέλευση του κοσυφοπεδίου. Επίσης θα πρέπει να πω ότι αυτή η ποσόστοση ακόμη δεν έχει εξαντληθεί, άρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Πάντως τυπικά προβλέπεται αυτό και βλέπουμε επίσης ότι και στην κυβέρνηση και σε άλλες κέρυες θέσεις ε, γυναίκες με τα απαραίτητα προσόντα κατέχουν τις θέσεις αυτές. Τώρα για τις εκλογές πρώτα απ' όλα. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτό που είπατε, για τη σημασία δηλαδή των εκλογών και την πρότασή σας. Κάποια μέλη της Επιτροπής Ετούτης εδώ και του Κοινοβουλίου γενικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αξιοποιήσουν τις επαφές που έχουν για να ενθαρρύνουν και τους Σέρβους Κοσοβάρους ως κοινότητα και το Βελιγράδι να συμμετάσχουν στις εκλογές. Πολύ θα το εκτιμούσα βέβαια, δεν χρειάζεται να σας το κρύψω θα εκτιμούσα όλη τη βοήθεια που μπορείτε να δώσετε. Τώρα, για ε, τη θέση μου, όπως είπα ήδη, τη ε, δυνατότητα αλληλεπίδρασης των δύο κοινοτήτων, την βλέπω. Επίσης πρέπει να πω ότι καμιά φορά δημιουργείται κάποια ε, σύγχυση αλλά και η εκπρόσωποι μου, ένας που ε, ανάλογα με τις αποστολές, ε, νομικό καθεστώς και εκλογές και εμείς θέλουμε να τα κρατήσουμε ξέχωρα. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο και είναι ευαίσθητα σε αυτό το θέμα, το σέβομαι απόλυτα, αλλά όλα τα κράτη-μέλη, να το πω και αυτό, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση του κυρίου Χουντή, Όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει να οριστεί ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κωσυφοπαίδιο και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια ευκαιρία αλλά και μια δυνατότητα για την περαιτέρω ε, ενίσχυση της σταθερότητας σε μια περιοχή όπου η χώρα σας, η Ελλάδα, ε, είναι σε ασθενή γειτονία και μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε σειρά θεμάτων που σε τελευταία ανάλυση θα αποβούν επωφελή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Παρά τα όσα είπα ήδη, ε, προσθέτω καταρχήν ότι ο συντονισμός μεταξύ της ε, παρουσίας του ΝΑΤΟ, της K4 και της ULEX ε, προχωρεί πολύ ικανοποιητικά. Ίσως γνωρίζετε ότι αν υπάρξει πρόβλημα σε πολιτικό επίπεδο προβλέπονται τρεις φάσεις. Το ένα είναι η τοπική αστυνομία να είναι η πρώτη που θα αντιδράσει. Κατά δεύτερο λόγο θα αντιδράσει η ULEX και κατά τρίτο λόγο θα παρέμβει η K4. Οπότε αν υπάρξει κάποια κοινωνική ταραχή, πάντα υπάρχει δυνατότητα ε, υποστηρικτικής παρέμβασης της K4. Όπως είπα ήδη, νομίζω ότι αποτελεί δείγμα ε, εμπιστοσύνη στην αυξανόμενη οριμότητα ε, της, των, των θεσμών εκεί που δείχνει ότι η K4 μπορεί να μειώσει τον αριθμό των στρατιωτών. Είμαστε στις 14.000 τότε και όλοι γνωρίζουμε τις γενικότερες προτεραιότητες. Η ιεράρχηση λοιπόν των αναγκών από τον ΝΑΤΟ φαίνεται να δικαιολογείται. Η παρουσία της Γιούλεξ δεν ε, είναι για την εκπαίδευση ή κατάρτιση πρωταρχικά. Αυτό έγινε επί δίκησης Ηνωμένων Εθνών τους προηγούμενους μήνες. Και είχε και επιτυχία αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οπότε ήδη η αστυνομία έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ε, επαγγελματισμού και αρτιότητας ε, ε, πολύ υψηλά. Αλλά αυτό που χρειάζεται ακόμα είναι αυτό που είπατε και εσείς, συμβουλευτικές υπηρεσίες, που θα, δηλαδή η συνοδεία των αστυνομικών κατά τα, την άσκηση των καθηκόντων τους, παρακολούθηση του τι γίνεται στα αστυνομικά τμήματα κλπ. Ο στόχος σε τελευταία ανάλυση, και εδώ σημειώνεται πρόοδος, ο απότερος στόχος είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τον πολυεθνικό χαρακτήρα της ε, αστυνομίας του Κωσόβου και όσο περισσότεροι Σέρβοι μπουν θα είναι καλό. Αυτό σημαίνει αυτό. Γιατί κάποια περίοδο έφευγαν οι Σέρβοι αστυνομικοί για πολιτικούς λόγους. Επιστρέφουν όμως. Πιστεύουμε ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης ε, για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μειοψηφουσών κοινοτήτων, των μειονοτήτων, ε, όσο γίνεται περισσότερη. γιατί θέλω να πω ότι η σύνθεση του προσωπικού της αστυνομίας ε, του Κωσυφοπεδίου πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο πολυεθνική. Δεν θέλω να να από πόσο θα διαρκέσει η αποστολή Ulex. Ε, υπάρχουν κάποιοι πόροι ε, σημαντικοί που υπάρχουν, αλλά καταρχήν ως θέμα αρχής θα ήθελα η διεθνής παρουσία ε, να μην κάνει αρμενική βίζητα θα λέγαμε, να μην ε, μείνει περισσότερο όσο χρειάζεται. Αλλά ίσως διαφορά το θέμα του κράτους δικαίου πρέπει να γίνει πάρα πολλή δουλειά ακόμα και νομίζω ότι είναι υποφελή όλων των κρατών μελών της Ένωσης να ε, θεωρηθεί το κράτος δικαίου ως μεγάλη προτεραιότητα. Δηλαδή να φροντίσουμε πριν φύγουμε να έχει πλήρως εγκαθιδρυθεί, θεσμοθετηθεί, ε, όχι ε, μόνο ως ε, προϊόν εξωτερικής επένδυσης, ούτως ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά η χώρα. Επανέρχομαι στις ερωτήσεις του κυρίου Χουντή. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το καθεστώς του κοσυφοπεδίου, δεν το έχουν αναγνωρίσει όλοι, αλλά όπως είπα υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι ε, που βρίσκουν σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη για το κοσυφοπέδιο και το τι πρέπει να γίνει εκεί. Και εδώ επάνω ε, γίνονται πρόοδοι και θεωρώ ότι θα συνεχίσει αυτή η καλή εξέλιξη με την υποστήριξη όλων των κρατών μελών. Δεν θέλω να ε, κάνω εικασίες σε σχέση με το μέλλον του καθεστώτος του κοσοϊφοπεδίου. Άλλοι, άλλοι έχουν πει ότι η ανεξαρτησία του κοσυφοπεδίου είναι μία αναστρέψιμη και νομίζω ότι η δήλωση είναι σημαντική και έτσι το ενδεχόμενο μιας νέας ειρηνευτικής διαδικασίας και ένα νέο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν βλέπω τώρα να αποτελεί ε, μια σημαντική πιθανότητα, και συμφωνούμε όλοι ότι αν υπήρχε, είχε υπάρξει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας, το, η έκβαση θα ήταν καλύτερη. Όμως είναι λυπηρό το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Φάιντ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ειδικό απεσταλμένο για όσα μας ανέφερε. Ε, θεωρώ ότι πολλά από αυτά είναι θετικά. Δύο σημεία, ε, ε, σε δύο σημεία ήθελα ε, να σταθώ. Ποιο είναι το ποσοστό του πληθυσμού το οποίο έχει αποχωρήσει από τη χώρα και σε ποια κοινότητα ανήκει και το δεύτερο είναι αν εσείς ως απεσταλμένος έχετε επαφή με το Βελιγράδι κατευθείαν για τα ζητήματα αυτά που αφορούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές παραδείγματο χάρη γιατί ακούστηκε ότι υπάρχουν φήμες ότι αποθαρρύνει η κυβέρνηση του Βελιγραδίου κάτι τέτοιο. Ε, αυτό είναι μια φήμη ή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή έχουν γίνει προσπάθειες προς την πλευρά του Βελιγραδίου για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των Σέρβων αφού και ο ίδιος είπατε ότι και σε επίπεδο αστυνομίας επιστρέφουν οι Σέρβοι και ότι κατά κάποιο τρόπο αρχίζουν να υπάρχουν κάποιες τοπικές ισορροπίες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Γιαννάκου. Ο συνάδελφος Τάλλερ έχει το λόγο. Rad bi vam čestitev, gospod Fajt, za vaše dobro upravljanje dela v nelahkih okoliščinah. Όπως ε, είπαν και οι προαλλαλήσαντες, οι εργασίες σας βαίνουν καλώς σε μια πλαισίωση που δεν είναι και τόσο καλή πάντα. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ για τα πολύ καλά αποτελέσματα. Στην πρώην Ιουκοσλαβία αυτά που είδαμε μας υπενθυμίζει την διάλυση των Δυτικών Αλφανίων, ε, Βαλκανίων που τότε αναφέραμε ως ε, Ιουκοσλαβία. Αυτό είδαμε και στο Κωσυφοπαίδιο. Είδαμε την κατάλυση της αυτονομίας και ε, αυτοκυριαρχίας από πλευράς Σέρβων και βλέπουμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία σταθεροποίηση στο κοσυφοπέδιο. Θα ήθελα να υποβάλω ε, μία ε, ερώτηση. Αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται ένα καθεστώς θεωρήσεων στην περιφέρεια και για την απελευθέρωση ε, των θεωρήσεων για τους κατοίκους της Μακεδονίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει την κατάσταση, διότι δεν θα απελευθερωθεί το καθεστώς θεωρήσεων για όλους τους πολίτες της ε, περιοχής θα δημιουργήσει μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ε, και δυσχέρειες για την χορήγηση διαβατηρίου στους πολίτες. Και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη Βοσνία Ερσεγοβίνη. Καθώς και στο κοσυφοπέδιο. Ποια είναι η γνώμη σας επί του θέματος. Ποιες είναι οι προοπτικές του κοσυφοπεδίου σε σχέση με το καθεστώς των θεωρήσεων, όπως προβλέπετε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ως κράτη-μέλη για την απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και για το κοσιφοπέδιο; Εσείς προβλέπετε κρατικές ενισχύσεις ως εμπειρογνώμων ή ηλική βοήθεια γενικά για την χορήγηση διαβατηρίων. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάλερ. Ο κύριος Σαρλάκη έχει το λόγο. Grazie Presidente. Uh, I appreciate uh, ε, Mr. Fate coming here. Εκτιμώ το ότι ο κύριος Φέιτ ήρθε εδώ για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό του κοσυφοπεδίου, να μας περιγράψει την κατάσταση και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή. Και Έχω πλήρη συνείδηση της δυσκολίας του έργου σας, διότι έχετε να κάνετε εκεί με τεράστια προβλήματα. Αλλά πρέπει να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένο από την εικόνα που μας δώσατε της κατάστασης. Η περισσότερη δήλωσή σας εστιάστηκε γύρω στις εκλογές, ε, ε, στην οικοδόμηση των θεσμικών οργάνων ε, και μιλήσατε μόνο επιφανειακά για μερικά θέματα ε, μεγάλης σημασίας για το Κωσυφοπαίδιο. Ε, μπορέσαμε να ασχοληθούμε, μπόρεσα να ασχοληθώ πριν μερικά χρόνια με το θέμα εργαζόμενος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Κωσυφοπαίδιο, εκτός βεβαίως από τις εθνοτικές εντάσεις και τις συνέπειες του πολέμου, είναι η τεράστια πολιτική διαφθορά το, το οργανωμένο έγκλημα, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η σωματεμπορία, η λαθρέα διακίνηση ανθρώπων, όλα αυτά αποτελούν σοβαρή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από την απειλή για τους Κωσοβάρους, η σχέση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και πολιτικής είναι βαθύτατη από τις πιο βαθιές που ξέρω η ε, δύναμη των ε, συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να συγκριθεί και είναι ακόμα μεγαλύτερη απειλή από τους ε, μεγάλους που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η, ανάμεσα στην Ιταλική μαφία και στην μαφία του, του Κωσυφοπέδιου θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μαφία του Κωσυφοπεδίου είναι πιο οργανωμένη, πιο ισχυρή ε, και η Σικελία είναι δυόμιση φορές το μέγεθος του Κωσυφοπεδίου. Διαρωτώ με ποιες είναι οι παράμετροι που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την επιτυχία ή αποτυχία της παρέμβασης σε μια χώρα. Αλλά στο Κωσυφοπέδιο θα έλεγα ότι παίρνοντας μόνον ε, το θέμα των εκλογών, αυτό λοιπόν που φαίνεται αμέσως ε, στην ζωή είναι βεβαίως μια παράμετρο σταθερότητας, αλλά δεν αρκεί. Βεβαίως είπατε ότι δεν είσαστε υπεύθυνο για τη δίκηση της χώρας, δεν είσαστε επικεφαλής της Γιούλεξ, είσαστε απλώ εκπρόσωπος, αλλά εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να παίξετε ένα ρόλο θέτοντας προτεραιότητες και θα ήθελα να μάθω για αυτές τις παραμέτρους για να δούμε εάν πράγματι προοδεύει το κοσυφοπέδιο στην πραγματικότητα. Ποιες είναι αυτές οι παράμετροι η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Είναι κέντρο όπου ξεπλένεται πάρα πολύ χρήμα, μαύρο χρήμα. Ε, δεν είναι μια χώρα με την πραγματική έννοια της λέξης. Δεν έχει γίνει ακόμα ε, δεκτή ε, στην διεθνή κοινότητα ως αξιόπιστος εταίρος και αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος αυτό, για τον οποίο δεν δίνονται θεωρήσεις στους Κωσοβάρους. Ίσως δεν μας αρέσει που το λέμε αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικότερος λόγος ότι όλες ε, οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν θέλουν να δοθεί θεώρηση στους Κωσοβάρους ε, διότι υπάρχει το ξέπλυμα χρήματος, ε, υπάρχουν, υπάρχει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το κοσυφοπαίδιο είναι απειλή για τις γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα κλπ θέλω να είμαι σύντομα ότι η αποστολή κοστίζει 260 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο η αποστολή Ulex. Ποιε είναι οι παράμετροι για να προσδιορίσουμε την επιτυχία ή αποτυχία. Μπορείτε να μας δώσετε μερικά στοιχεία για τα όσα γνωρίζετε για την κατάσταση, για αυτά που νομίζω ότι είναι οι πραγματικές παράμετροι επιτυχίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο και δίνω το λόγο στον κύριο Κουμουτσάκο. Ε, ε ευχαριστώ πολύ τον ε, ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενημέρωση που μας έκανε για την πορεία του πράγματι δύσκολου και σύνθετου έργου και της αποστολής που έχει η Ιούλεξ στο Κόσοβο. Θα ήθελα ε, να ρωτήσω κάτι που αφορά περισσότερο τον πολιτικό περίγυρο και πώς αυτός μπορεί να επηρεάσει την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα <clears throat> τις πολιτικές εξελίξεις στο κόσμο. Συγκεκριμένα αναφέρομαι, όπως ξέρετε, στο γεγονός ότι το Βελιγράδι έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προκειμένου το δικαστήριο να γνωμοδοτήσει εάν η ανακήρυξη, η μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας του Κωσόβου ήταν νόμιμη ή όχι. Αυτή τη στιγμή ακόμα η γνωμοδότηση δεν έχει βγει. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον ε, κύριο Φέιθ αν υπάρχει κάποια εκτίμηση στο πότε θα εκδοθεί η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Ε, επαναλαμβάνω, γιατί ίσως δεν με ακούγατε, ε, αν έχετε κάποια εκτίμηση κύριε Φέιθ για το πότε θα εκδοθεί αυτή η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και πώς αυτή η γνωμοδότηση θα μπορούσε να επηρεάσει το γενικό πολιτικό κλίμα στο Κόσοβο. Ειδικά εάν η γνωμοδότηση αυτή εκδοθεί πριν από την δεξιαγωγή των κρίσιμων τοπικών εκλογών του Νοεμβρίου. Και βεβαίως είναι προφανές ότι ανάλογα με το περιεχόμενο αυτής της γνωμοδότησης θα υπάρχει και η ανάλογη επίδραση. Αν η γνωμοδότηση αυτή δείχνει περισσότερο προς το ότι ήταν απόλυτα νόμιμη η ανεξαρτησία, αυτό θα έχει ένα αλφα αντίκτυπο. Εάν όμω η γνωμοδότηση κινηθεί προ την κατεύθυνση τη μη νόμιμη ανακήρυξη ανεξαρτησία. αυτό είναι βέβαιο ότι θα έχει έναν τελείω διαφορετικό αντίκτυπο και για τι εκλογέ, αλλά ενδεχομένω και για την αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κόσοβο. Θα ήθελα σα παρακαλώ πάρα πολύ να έχω τι σκέψει και τι εκτιμήσει σα για αυτά τα ζητήματα που είναι αρκετά σημαντικά πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουμουτσάκο. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκόμες και έτσι θα έχουμε πέντε παρεμβαίνοντας. Και μετά θα απαντήσω ο Δόκτωρ Φάιτ. Η κυρία Γκόμες, με συγχωρείτε. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, που ξαναβλέπω τον ειδικό απεσταλμένο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Για να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα και την διαφθορά, θα πρέπει να υπάρχει οικονομική σταθερότητα στο Κωσυφοπέδιο Και αυτός είναι ένας τομέας όπου η Ευρώπη απέτυχε κατά τον, τον επιμερισμό ε, καθηκόντων από την ΑΝΜΕΚ. Υπάρχουν ε, οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Μιλήσαμε για μία νέα ε, υδροηλεκτρική μονάδα. Οι γυναίκες, εκτός από το γεγονός ότι αποτελούν αντικείμενο ε, σωματεμπορίας, η Ιούλεξ προβλέπει μία ε, μονάδα και για αυτές, δηλαδή για τις γυναίκες της, ε, του Κωσυφοπεδίου και τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας θέσω το ερώτημα των πρέσβεων. δεν υπάρχει καμία πρέσβης γυναίκα από το κοσυφοπέδιο. Έχει αλλάξει η κατάσταση έκτοτε. Θα μπορείτε, θα μπορούσατε να μου πείτε πώς έχει κατάσταση της Γιούλεξ στη Μητροβίτσα. Πώς ε, λειτουργεί. Λειτουργεί αυτό το δικαστήριο. Και τέλος η Γιούλεξ ε, χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη σε επίπεδο εισαγγελέων. Αυτό γιατί δεν προωθείται, σχετίζεται με μια ενδεχόμενη χρηματοδότηση, είναι άλλοι λόγοι. Ε, Πριν να ε, δώσω το λόγο στο δόκτορα Φέιτ θα ήθελα να απαντήσω στο τελευταίο ερώτημα της κυρίας Γκόμες. Η συνάδελφος Νέιτς υπέβαλε μία τροπολογία στο σχέδιο προϋπολογισμού που προβλέπει ένα ειδικό κονδύλιο για να βοηθήσουμε την γυναικεία παρουσία στα πλαίσια των ειδικών αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αντιμετώπιση σεναρίων κρίσης. Άρα ε, έχει αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δόκτωρα Φάιτ, έχετε το λόγο. Για να αρχίσω, πρώτα απ' όλα από την ερώτηση της κυρίας Γιαννάκου. Μετά τις βιότητες, στο τέλος της δεκαετίας ε, του 90, 98, 99, πάρα πολλοί Σέρβοι και ακόμα και το 2000-2001 πάρα πολλοί ε, Σέρβοι έφυγαν από το Κωσυφοπέδιο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη προτεραιότητα για μένα να ενθαρρύνω την επιστροφή των Σέρβων στις πατροχονικές τους εστίες στο Κωσυφοπέδιο. Και ε, ε, σκέφτηκα διάφορα μέτρα ούτως ώστε να μπορέσουν οι Σέρβοι ε, να εξακολουθήσουν να έχουν ασφαλή διαβίωση στο κοσυφοπέδιο. Πρέπει να πω ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την επιστροφή είναι περιορισμένα και ότι χρειάζεται να αυξηθούν με βοήθεια διαφόρων οργανώσεων εγώ προσωπικά δεν έχω το προνόμιο να είμαι σε επαφή με το Βελιγράδι για το θέμα αυτό. Είμαι βεβαίως διαθέσιμος. Προσπαθούμε να επιταχύνουμε την διαδικασία επαναπατρισμού, επανόδου. Υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν επιστρέψει και νομίζουμε ότι θα πρέπει να καταστεί δυνατόν, δεν είναι μόνο ε, απαραίτητο, αλλά ότι θα πρέπει να καταστεί ε, δυνατός ο επαναπατρισμός ε, μεγαλύτερου όγκου ατόμων. Σχετικά με τις θεωρήσεις, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Τάλερ να μην προκαταλαμβάνουμε την παρουσίαση που θα κάνει ο Επίτροπος αύριο εδώ, ο Επίτροπος Ρέιν σχετικά ε, με την ελευθεροποίηση των θεωρήσεων. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για τη χώρα είναι να έχουν ε, την θεσμική ικανότητα ούτως ώστε να μπορούν να έχουν ένα περιβάλλον όπου ελεύθερα ε, θα μπορούν να δίνονται θεωρήσεις, όπου θα είναι ασφαλή τα σύνορα ούτε ώστε να έχουν την ελευθερία οι πολίτες της χώρας. Στην περίπτωση του Κωσυφοπεδίου, δεν υπάρχουν βιομετρικά διαβατήρια στο Κωσυφοπέδιο, θα μπορούσαν να εισαχθούν σύντομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμέσου της Ιούλεξ προσπαθεί ε, να εισαγάγει ε, διάφορα μέσα ούτως ώστε να καταστεί δυνατή συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο για θέματα αστυνομίας και τελωνίων που είναι απαιτήσει τώρα, που είναι κριτήρια ούτως ώστε το κοσυφοπέδιο να μπορέσει να επιτύχει αυτήν την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ελέγχθηκε επίσης από τον Χαβιέ Σολάνα ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία και ελπίζουμε με την πάροδο του χρόνου θα έρθει η κατάλληλη στιγμή ούτω ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό, ούτω ώστε να έχουμε, όπως είπατε και εσείς, μια περιοχή όπου δεν θα χρειάζονται πουθενά θεωρήσεις. Σημείωσα με μεγάλο ενδιαφέρον την περιγραφή του κυρίου Αλάτσι σχετικά με την σοβαρότητα των προβλημάτων δεν νομίζω ότι τα όσα είπα έρχονται σε αντίφαση με τα όσα είπατε εσείς. Πρόκειται για σοβαρά προβλήματα. Και είναι ο λόγος για τον οποίο συμφωνήσαμε να αναπτύξουμε την μεγαλύτερη αποστολή ΕΠΑΑ, την μη στρατιωτική, εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ποια θα είναι το τελικό στάδιο και ποιες είναι οι παράμετροι που θα προσδιορίσουν την επιτυχία. Καμιά φορά μια αποστολή αλλάζει, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με το κοσυφοπέδιο θα πρέπει να έχουμε μια ποιότητα του κράτους δικαίου που θα επιτρέψει στο κοσυφοπέδιο μια μέρα ε, να φτάσει πιο κοντά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχουμε βεβαίως κάποια επιρροή πάνω στις αρχές του κοσυφοπεδίου, ούτω ώστε να συνεργάζονται καλά με την αποστολή Γιούλεξ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και συμφέρον, όπως ξέρετε, για το λαό του Κωσυφοπεδίου να γίνει μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Γι' αυτό οι ηγέτες, οι αρχές βρίσκονται υποπίεση για να επιδείξουν πρόοδο. Είναι αληθές, μίλησα για την οικοδόμηση των θεσμών, αλλά η επόμενη φάση θα εστιαστεί πολύ περισσότερο για το πώς θα λειτουργήσουν αυτά τα θεσμικά όργανα σύμφωνα με τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς και τους διεθνείς. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με θέματα διακυβέρνησης, με θέματα λογοδοσίας και θα πρέπει να καταπολεμηθούν περιπτώσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Για αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία ή να σας πω, να σας δώσω ενδείξεις για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η καταπολέμηση και αυτός ο αγώνας πως θα γίνουν ορισμένες έρευνες. Αλλά μπορώ να πω ότι υπάρχει προσδοκία στο Κωσυφοπέδιο, κυρίως μεταξύ των πολιτών του Κωσυφοπεδίου, ότι η Ιούλεξ, η αποστολή Ιούλεξ μπορεί να επιτύχει ορισμένες ε, περιπτώσεις, ορισμένα άτομα, ε, εγκληματικά στοιχεία να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Ούτω ώστε να καταπομιλεμηθεί η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι η Επίτροπη ότι ενδιαφέρεται πολύ για τα θέματα αυτά η Κομισιό παραμετός χάρη για τους δημόσιους διαγωνισμούς, για τα δημόσια έργα όπου υπάρχει ε, μεγάλος κίνδυνος κακών πρακτικών ε, για αυτά τα θέματα ασχολούμεθα εντατικά. Τώρα περνάω στις ερωτήσεις που έθεσε ο κύριος Κουμουτσάκος σχετικά με το Διεθνές Δικαστήριο. Δεν μπορώ, ε, δεν μπορώ εγώ να προβλέψω ποια θα είναι η γνωμοδότηση του δικαστηρίου. Μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις αλλά δεν θα είναι αυτό πάρα πολύ παραγωγικό. Αυτό που μπορώ να σας πω με κάποια εμπιστοσύνη είναι ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος, πολύ περισσότερος χρόνος από μέχρι τον Νοέμβριο. Ξέρουμε ότι το δικαστήριο θα οργανώσει ακροάσεις το Δεκέμβριο, προφορικές ακροάσεις και μετά οι δικαστές θα αρχίσουν να εργάζονται για τα συμπεράσματα, για τη γνωμοδότηση και ελπίζουμε ότι ε, η γνωμοδότηση αυτή ε, θα, ε, θα υπάρξει στα μέσα. Ε, δεν πρόκειται για μια απόφαση, αλλά πρόκειται για μια γνωμοδότηση που θα έχουμε, ελπίζω, στα μέσα του επομένου έτους. Συμβουλευτική γνωμοδότηση που δεν θα είναι δεσμευτική για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπέδιο βεβαίως θα είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει τα ίδια τα κράτη αυτά να κρίνουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, οι επιπτώσεις ε, της συμβουλευτικής γνωμοδότησης. Έφτασα τώρα στην κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια, κυρία μου. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι η οικονομική κατάσταση στο Πέδιο... είναι ακόμη πολύ εύθραυστη διότι η οικονομική κρίση είχε επιπτώσεις και οι επιπτώσεις αυτές αυξάνονται τώρα και έχουμε τώρα μερικές άλλες παρενέργειες διότι το Κωσυφοπέδιο έχει μια υπανάπτυκτη οικονομία που δεν είναι καλά ενσωματωμένη στην παγκόσμια οικονομία και γι' αυτό χρειάστηκε πιο πολύ χρόνος οι διακλαδώσεις της οικονομική παγκόσμια κρίσης να φτάσουν στο κοσυφοπέδιο. Αλλά έχουμε τραγικές συνέπειες πάνω στην απασχόληση και στις ξένες επενδύσεις. Επίσης, το θέμα που έχει σημασία είναι η ιδιωτικοποίηση, αναφερθήκατε στον τομέα της ενέργειας Υπάρχουν μερικές πηγές εξαγωγών, αν τα πράγματα ε, εξελιχθούν καλά, υπάρχουν ορισμένες, ε, υπάρχει λιγνίτης και το προϊόν αυτόν ε, μπορεί να προμηθεύσει ηλεκτρισμό στην περιοχή. Αλλά η διαδικασία ιδιωτικοποίησης επηρεάστηκε από μία ή δύο αποσύρσεις δυνητικών ενδιαφερομένων για αυτό το, το νόμιλο και σύνεπώς θα πρέπει να αποφασιστεί ε, η μελλοντική διαδρομή προσεχώς. Ελπίζω να ληφθεί μια απόφαση και να υπάρξουν συναλλαγές ή αλλιώς ο ηλεκτρισμός θα πρέπει να εισάγεται με ηλεκτρική ενέργεια με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Έχουμε βεβαίως θέσεις που καλύπτονται από γυναίκες. Η υφυπουργό του Κωσυφοπεδίου για τα εξωτερικά θέματα ασκεί το λειτουργήμά της με μεγάλο επαγγελματισμό σχετικά με τη Μητροβίτσα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο σημείο όπου ε, Σερβοί και οι Αλβανοί του Κωσυφοπεδίου, οι ε, δικαστές ε, και οι εισαγγελείς να έχουν αρχίσει να εργάζονται και να έχουν επαφές με τους ομολόγους τους στο βορρά με το Βελιγράδι. Ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα. Και θα ήθελα να πω στο τέλος και εδώ ίσως να χρειάζομαι και τη βοήθεια της Επιτροπής επίσης και επανέρχομαι στα όσα είπε ο κύριος Σαλάτσια σχετικά με την σοβαρότητα του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ίσως να χρειαζόμαστε περισσότερους εισαγγελείς. Ίσως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν περισσότερους εισαγγελείς για να λάβουν τις σοβαρές υποθέσεις και περιπτώσεις. Είναι βεβαίως δυνατόν να κάνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη για μια τέτοια βοήθεια, για εμπειρογνώμονες, ούτω ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία για την αποστολή Ιούλεξ. Ευχαριστούμε, δόκτωρα Φάιντ. Η παρέμβασή σας ήταν για μια φορά ε, ακριβής και στόχοθετημένη. Ας περάσουμε στους τελευταίους πέντε συναδέλφους. Και αρχίζουμε τον κύριο Χάουιτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Φέιτ που ήρθατε σήμερα. Το Κοινοβούλιο στηρίζει ιδιαίτερα το έργο σας, το ξέρετε, ευχόμεθα κάθε επιτυχία. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, ε, διαδηλώνουμε και, διαδηλώνω και εγώ το ενδιαφέρον μας για την παρακολούθηση των εκλογών, όχι μόνο στα πλαίσια ε, των ευρωπαϊκών θεμάτων, αλλά χάρη στον εκδημοκρατισμό σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία στις ε, αποστολές ε, παρακολούθησης εκλογών. Τώρα, για τις ερωτήσεις μου. Η θητεία σας βεβαίως περιλαμβάνει στήριξη και σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών, ελευθεριών. Και ερωτώ, Πώς κρίνεται, ποιες κρίνεται να είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις στον τομέα αυτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στο Κωσυφοπαίδιο. Δεύτερον, Ακούσαμε τα σχόλιά σας σε σχέση με την υποστήριξη ε, από τη διεθνή παρουσία. Αλλά ε, υπάρχουν κάποιες τάσεις ή διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν, γιατί δεν ε, είναι μόνο θέμα που περιορίζεται στο κοσυφοπέδιο, αλλά οπουδήποτε υπάρχουν διεθνείς δυνάμεις σε περιοχές κρίσεων και συγκρούσεων. Ε, καλό θα είναι να ακούσουμε σε αυτό το πλαίσιο τα σχόλιά σας, λοιπόν. Τέλος, ε, σας άκουσα... Ε, όταν μιλήσατε για την ε, παλινόστηση των προσφύγων, την συνεργασία τελωνίων, αστυνομιών κλπ. Μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση της κατάστασης της σημερινής σε σχέση με το πώς ήταν πριν από ένα χρόνο για να δούμε ας πούμε τι ε, διμερείς ε, εξελίξεις σημειώθηκαν μεταξύ Παιδίου και γειτονικών χωρών. Ευχαριστούμε κύριε Χάουιτ. Ο κύριος Βαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα στον κύριο Φάιτ. Γράφει στην έκθεσή του ότι η πολιτική των Σέρβων έγκυται στην ε, ε, εξασφάλιση των δημοσίων υπηρεσιών στους θυλάκους αυτούς που θα πρέπει να είναι υπό την αιγίδα του ε, Βελιγραδίου. αυτή την έννοια είναι δύσκολο να υπάρξει επιτόπιος έλεγχος. Αυτή τη στιγμή είναι δυνατόν να σταματήσουμε αυτό τον σερβικό έλεγχο και τι έχει γίνει από αυτού. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Βαμπάλεν. Η συνάδελφος Κύριλοφ έχει το λόγο. Στο Ο συνάδελφος Κύριλοφ. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Ε, συμφωνώ με τον κύριο Αλάτσι, τον συνάδελφο Αλάτσι. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του απόλυτα και είμαι ευτυχής που ο κύριος ε, Φέιθ ε, έχει κάποια γνώση της κατάστασης. Επιπροσθέτως ανησυχώ και για κάτι ακόμα. Δηλαδή, όλη αυτή την κατάσταση με τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα και σε ποιο βαθμό μπορεί ε, η μελλοντική εξέλιξη να επηρεαστεί από τους πολιτικούς ε, γιατί η κυρία Σφέιθ γνωρίζει πολύ καλά νομίζω ότι το οργανωμένο έγκλημα διεισδύει παντού ακόμα και στο επίπεδο των κορυφαίων πολιτικών του Κωσόβου. Η πρόκληση είναι μεγάλη αν λοιπόν δεν μας απασχολήσει όπως πρέπει και όσο πρέπει, μπορεί να βρεθούμε προ σοβαροτά της ε, καταστάσεως. Γέλασα λίγο με το πώς χρησιμοποιήσατε την λέξη mentoring, παροχή με συμβουλευτικών υπηρεσιών, ρόλο μέντορα. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα βοηθήσει αυτό το mentoring στο μέλλον. Αρκεί Μιλάτε για διώξεις. Πώς θα, οι, οι, οι διώκοντες θα δράσουν. Γιατί από νομικής πλευράς είναι ολισθηρό το έδαφος. Ας φανταστούμε ας πούμε ότι αρχίζει να γίνεται μια ε, μάχη που θα πλήξει πολλούς κύκλους. Τελευταία ακούω πολλά για την ε, αυτοδιάθεση του κοσυφοπεδίου και ομολογώ ότι πιστεύω ότι αυτό δεν είναι κάτι που απορρέει από την κοινωνία των πολιτών, από τους πολίτες εκεί. Μπορεί στο τέλος να φτάσουμε σε μια κατάσταση, το απέφχομαι και σας εύχομαι σας κάθε επιτυχία, αλλά μπορεί ας πούμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε ένα στάδιο όπου η μάχη αυτή θα γίνει πιο έντονη, αποτελεσματική και θα δούμε τι ε, επιπτώσεις θα έχει γενικότερα. Αυτή η ιονή κοινωνία, γιατί ε, κάποιοι θα θυμούνται ίσως ότι η ανεξαρτησία ήταν επιθυμητή από διαφορετικούς κύκλους για διαφορετικούς λόγους. Ας πούμε λοιπόν ότι φτάνει ένα σημείο, ε, φτάνουν σε ένα σημείο και λένε δεν σας θέλουμε πια εσάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρουσία σας. Ήδη φαίνεται αυτό από την, ε, ε, τους στόχους, της, ορισμένους στόχους της αυτοδιάθεσης. Εννοώ ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρό πρόβλημα αν δεν μελετήσουμε σε βάθος το πρόβλημα. Ε, αυτό Ίσως είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε με τα τελωνία. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και εδώ αλλά ξέρουμε πολύ καλά το παράνομο εμπόριο από τι κανάλια περνάει. Δεν είναι δύο σημεία μόνο. Περνάνε τα βουνά από παντού, από κάθε σημείο. Δεν θέλω να σας αποθαρρύνω προς Θεού. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που το κάνουν. Αλλά εδώ πόρο απέχομαι από την επίτευξη των στόχων. Πρέπει να πιο ρεαλιστικά να την αξιολογήσουμε και να την εκτιμήσουμε. Αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, ολόψυχα εύχομαι επιτυχία σε εσά. Ο συνάδελφος Κάτσιν έχει το Grazie Presidente Albertini. Gospod Fejt, nisem zadovoljen z vašimi odgovori, ko gre za vizni režim. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις ε, απαντήσεις σας σε σχέση με το καθεστώς των θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε πολλά λάθη στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι Ούγγροι της Σερβίας προτιμούν την Ουγγρική υπηκότητα, οι Βούλγαροι στη Μακεδονία τη Βουλγαρική υπηκότητα και ούτω καθεξής. Και τώρα οι Σέρβοι, οι οποίοι διαμένουν στο Κωσυφοπέδιο, θα προτιμήσουν την Σερβική υπηκότητα. Άρα στην ουσία διχάζεται του Σέρβους, δηλαδή στους Σέρβους, τους κανονικούς Σέρβους, τους πραγματικούς Σέρβους και στους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Ε, προβαίνεται εδώ σε μία διάκριση, κάτι το οποίο ε, θα οδηγήσει τους Σέρβους να απομακρυνθούν από το Κωσυφοπέδιο και να μεταβούν στη Σερβία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Η μόνη λύση έμπρακτα για τους ε, κατοίκους του Κωσυφοπεδίου θα είναι το οργανωμένο ε, έγκλημα. Τώρα, ως προς τα βιομετρικά διαβατήρια, εγώ δεν έχω βιομετρικό, βιομετρικό διαβατήριο και νομίζω πολλοί μεταξύ ημών δεν διαθέτουν τέτοιο διαβατήριο. Αυτό δεν αποτελεί λύση κατά την άποψή μου. Τη στιγμή που δεν ε, διαθέτουμε μια πολιτική αρχών και δεν ξέρουμε πώς ε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους έτσι ώστε να θεωρήσουν ε, αυτούς επιθυμητούς και να έχουν ίσα δικαιώματα, τότε δεν καταφέρνουμε τίποτα. Πώς θα δράσετε, τι θα προτείνετε στην Επιτροπή σύμφωνα με την ε, πείρα της EULEX, έτσι ώστε να αλλάξει η πολιτική θεωρήσεων στο κοσυφοπέδιο δεν υπήρχε... Ε, ε, Ευχαριστούμε κύριε Κάτσιν. Η κυρία Μονιστή Κουίτσα. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Κάτσιν, δηλαδή τη στιγμή που δεν επεκτείνεται το καθεστώς των θεωρήσεων και στους ε, Σέρβους του Κωσυφοπεδίου θα τους εκδιώξει από το έδαφος. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάμε στον ε, πολυεθνοτικό χαρακτήρα δηλαδή. Στο γλωσσάρι που χρησιμοποιούμε και σε καμία δήλωση του ειδικού αντιπροσώπου δεν γίνεται καμία ε, μνήα εξωτερικών ε, σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν μιλάτε για εξωτερική νομιμότητα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι δραστηριότητες μας και στην ε, περιφέρεια αυτή. Και αυτό θα διευκόλυνε τη γενικότερη δράση μας στην περιφέρεια. Ευχαριστούμε. Και τώρα δίνω λόγο στον δόκτωρα Φάιτ για τις τελικές απαντήσεις. Ίσως σε αυτό το τελευταίο γύρο απαντήσεων θα πρέπει να πάω από το τέλος προς την αρχή και να διαβεβαιώσω την κυρία Μουνίζ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εργάζεται ε, πάνω στη βάση του διεθνούς δικαίου. Βέβαια, είναι λυπηρό ότι καμιά φορά υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες δικαίου. Τι είναι το διεθνές δίκαιο δηλαδή. Αλλά κατά τα άλλα επιβεβαιώνω ότι οτιδήποτε κάνουμε και όλες οι δράσεις μας στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και της ΕΠΑΑ συμπεριλαμβανομένων ε, των Αποστολών ε, για το κράτος δικαίου, ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κωσυφοπαίδιο, θεωρούμε ότι συνάδει 100% με το διεθνές δίκαιο. Και πάλι θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας για το γεγονός ότι πολλά θέματα που ε, τέθησαν για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων θα πρέπει να απαντηθούν από τον Επίτροπο, ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος να δώσει τα επιχειρήματα που αξιοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, υποβολή των προτάσεών της. Τώρα για το συγκεκριμένο ζήτημα των ε, Σέρβων Κωσοβάρων που όπως είπατε δεν ε, έπαιρναν θεώρηση, δεν τους έδιναν. Μπορείτε να το δείτε και αλλιώς. Αν η απόφαση επέκταση της απελευθέρωσης των θεωρήσεων είχε συμπεριλάβει τη σέρβικη κοινότητα στο κοσυφοπαίδιο, θα Αναρωτιόταν κανείς, οι επιπτώσεις δεν θα ήταν ότι οι Σέρβοι κοσοβαροι θα στρέφονταν περισσότερο προς το Βελιγράδι έτσι και θα ενδιαφέρονταν λιγότερο, πολύ λιγότερο για την ενσωμάτωση ε, με τους Αλβανούς κοσοβαρους στο Κοσυφοπέδιο Για να ισχύσει η απελευθέρωση των θεωρήσεων σε όλους τους κατοίκους του κοσυφοπεδίου και αυτό είναι προσωπική μου αντίληψη πιο καλό ε, η συμπερίληψη αυτή θα οδηγούσε σε ευκολότερη ενσωμάτωση από ότι μια διαφοροποίηση ε, με βάση τις διαφορετικές κοινότητες στο κοσυφοπέδιο. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το δείτε ως προσωπική μου ε, γνώμη και γι' αυτό θεωρώ ότι καλές είναι οι αποφάσεις που τυχόν ληφθούν ε, για την απελευθέρωση εφόσον όλοι οι κάτοικοι του κόσυφο ε, ε συμφωνώ με τις αποφάσεις σε σχέση με τις αποφάσεις ε, για την απελευθέρωση των θεωρήσεων ε, σε σχέση με τις διαφορετικές κοινότητες. Μπορώ να ε, κατανοήσω αυτό που είπε ο κύριος Κύριλοφ σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτικών σε εγκληματικές δραστηριότητες και στον κίνδυνο, αν η EULEX έχει επιτυχία, μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις ή κάποιο αρνητικό αντίκτυπο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όμως ε, εξακολουθώ να επιμένω και το λέω και προς άλλους συναδέλφους σας που είπαν κάτι παρόμοιο, υπάρχει πολύ ισχυρή ε, επιρροή, μόχλευση τώρα λόγω της ευρωπαϊκής ε, προοπτικής. Πολλοί κοσοβάροι πολιτικοί αλλά και πολίτες κοσοβάροι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή την προοπτική και τα ωφέλη από μια περαιτέρω ε, γυτνίαση και προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απελευθέρωση των θεωρήσεων είναι ένα θέμα. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει για πολλούς λόγους ακόμα, κυρίως τεχνικούς λόγους. Γιατί η συγκριτική αξιολόγηση, τα benchmark που ανέφερα και που θα τα εξηγήσει περισσότερο ο Επίτροπος Ρεν δεν έχουν ακόμη ε, υλοποιηθεί από το κοσυφοπέδιο. Όμως παραμένει σε μια διαδικασία η χώρα αυτή και η Κομισιόν θα διευκρινίσει τα περαιτέρω βήματα στα οποία θα προβεί στα Βαλκάνια και θα ακούσετε από τον Επίτροπο τι, ποια θα είναι αυτά. Όμως η η ελξιμότητα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσέγγιση ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κινητήρια δύναμη για το λαό και τους πολιτικούς του Κωσυφοπεδίου που θέλουν να ε, κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Θα έλεγα επίσης ε, ότι τους ενδιαφέρει να συνεργαστούν με την EULEX στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ίσως θεωρείτε ότι είμαι υπεραισιόδοξος, αλλά εγώ νομίζω ότι αν ε, δουλέψει κανείς σε τέτοια διαχείριση κρίσεων μετά από συγκρούσεις και δεν είναι ε, αισιόδοξο, τότε η ζωή θα γίνει έναν υπόφορο βάρος και δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Σε τελευταία ανάλυση νομίζω ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα κύριε Κύριλοφ και ας ελπίσουμε βέβαια ότι θα με περαιτέρω πρόοδο γιατί και η αποστολή Γιούλεξ στο κάτω-κάτω ε, άρχισε εδώ και 9 μήνες έτσι δεν είναι. Οπότε ακόμα, άρχισε ε, 9 μήνες πριν μόλις. Οπότε υπάρχει ακόμα περιθώριο για να βελτιωθεί και για να κριθεί ε, πιο εντελεχώς αλλά και πιο θετικά. Για τον κύριο Φον Μπάλεν, ε, μου φαίνεται ότι υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ μεταξύ μας. Εγώ ούτε το έγραψα ποτέ, ούτε το είπα ποτέ ότι είμαι υπέρ τη συμμετοχή των Σέρβων στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Κωσυφοπέδιο. Αυτό που είπα και αυτό που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι πολύ στο αντίθετο. Αλλά μιλάμε για ε, ε, ενισχυμένη αυτονομία ε, δικαιώματα αυτονομίας. Αυτό σημαίνει ότι η κοινότητα των Σέρβων αφενός θα δεχτεί να συνεργαστεί με την κεντρική διοίκηση Δεύτερον, θα υπάρχουν προνομιακοί δεσμοί στο μέλλον, και αυτό το συμφώνησαν οι αρχές της Πρίστινα, θα υπάρχουν προνομιακοί, προνομιακές, συνδέσεις σε ό,τι αφορά την ε, ε, ροή κεφαλαίων ούτως ώστε να ε, μπορούν να βοηθηθούν στους τομείς της υγείας, της παιδείας κλπ. Και ε, αυτά θα πρέπει να γίνονται υποκαθεστώς απόλυτης, αδια... διαφάνειας. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια ε, στο Πέδιο. Δεν είναι δηλαδή αυτό ένα άνοιγμα προς το Βελιγράδι ε, που θα κληθεί σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης να θέσει υπό τον έλεγχό του το Πέδιο προς Θεού είναι ένα χαρακτηριστικό ε, των ενισχυμένων δικαιωμάτων αυτονομίας που προσφέρονται στην Σέρβικη κοινότητα και ελπίζω πραγματικά ότι θα δράξει την ευκαιρία η κοινότητα των Σέρβων και θα συμφωνήσει και το Βελιγράδι ότι αυτό είναι ε, εποφελές για την κοινότητα των Σέρβων. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Χάουιτ που ε, ξέφρασε την υποστήριξή του και το ενδιαφέρον του για την παρακολούθηση των εκλογών και το ενδεχόμενο το Κοινοβούλιο να συμβάλλει ε, σε αυτό το θέμα. Η διεθνής παρουσία στο Κωσυφοπέδιο τα προηγούμενα χρόνια πάντοτε ε, ήταν θετική και πάντοτε γινόταν δεκτή θετικά από το τοπικό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η εντύπωση ότι αυτή η διεθνής ε, παρουσία ε, θεωρήθηκε θετική και όχι καταπιεστική. Ε, είχε πολλές επιτυχίες η παρουσία των Ηνωμένων Εθνών και έδωσε και καλά αποτελέσματα αφού βελτίωσε και ενίσχυσε το επίπεδο της διακυβέρνησης στη χώρα. Πριν από Υπήρξε όμως ε, μια βεβαιότητα για το καθεστώς που διαρκεί 9 χρόνια. Άρα κύριες αποφάσεις ε, δεν, δεν μπορούσαν να ληφθούν από τους ίδιους τους Κωσοβάρους. Από την αρχή θεώρησα και συμφωνεί και, η, και ο επικεφαλής της Γιούλεξ ε, είναι ότι τώρα πρέπει να υπογραμμίσουμε την τοπική ε, ε, ε, η κυριότητα. Οι σοβαροί πρέπει να πάρουν αποφάσεις, πάνω απ' όλα να αναλάβουν ευθύνη να λογοδοτούν για τα έργα τους. Αλλιώς θα χρειαστεί, φοβάμαι, να μείνουμε για πάρα πολύ μακρό χρονικό διάστημα στο κοσυφοπαίδιο και αντί να επιταχύνουμε θα επιβραδύνουμε την προορία της χώρας αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε τη σωστή τακτική θα έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία σε μικρότερο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσουμε εμείς τις ίδιες τις αρχές και τις δράσεις τους. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό και ελπίζω ότι θα ε, ε, βρω σύμφωνους και εσάς πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον δόκτορα Πάιτ, εξ ονόματος ε, όλων. Βεβαίως αυτό το κάνατε και με τις ε, μεμονωμένες σας παρεμβάσεις. Απλώς το επιβεβαιώνω σε αυτή την τελική φάση της συζήτησης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους διότι συνεισφέρατε σε αυτή τη συζήτηση με θέματα επικαιρότητα και ουσίας προβαίνοντας σε μία εις βάθος ανάλυση αυτής της επιμέρους θεματικές. Νομίζω ακούγοντας την κυρία Πακ, τον κύριο Σβόμποντα και άλλους και ακούγοντας και τα λόγα του δόκτωρος Φάιτ, φτάνουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και μπορούμε ανακεφαλαιώνοντας τη συζήτηση να πούμε ότι υπάρχει η συλλογική επιθυμία να αποστείλουμε μία αντιπροσωπεία ad hoc και που για οργανωτικούς λόγους ε, δεν μπορεί να είναι μια πραγματική αποστολή παρατηρητών σε σχέση με το, ως προς το εκλογικό σενάριο, θα δούμε πώς θα ορίσουμε την πλαισίωση αυτής της αντιπροσωπείας με τον Dr. Φάιτ. Μπορούμε λοιπόν να αποστείλουμε μια αντιπροσωπεία ε, που να απαρτίζεται από μέλη αυτής της Επιτροπής και με άλλους ε, αντιπροσώπους που ασχολούνται με τις όμορες περιοχές για να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα στείλω μία επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να προτείνω κάτι τέτοιο στην επόμενη ε, Επιτροπή στο επόμενο διαβριμένο Προεδρείο και στη διάσκεψη των Προέδρων για να οργανώσουμε ε, αυτή την πλαισίωση. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φάιτ, ο οποίος δέχτηκε αυτή τη συνάντηση. Γνωρίζει εις βάθος το όλο ζήτημα και γι' αυτό μπόρεσε να είναι τόσο αποδοτικός και αποτελεσματικός και να μας δώσει όλες τις πληροφορίες που ήταν χρήσιμες, απόλυτα χρήσιμες. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ξαναειδωθούμε σύντομα. Allora, ehm, Υπάρχουν και άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη που είχαν θυγεί αρχικά σε σχέση με το θέμα αυτό. Καταρχήν η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 16 Ιουλίου και 21 Ιουλίου 2009. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, από πλευρά συναδέλφων θεωρώ ότι εγκρίνονται. Νομίζω ότι εγκρίνονται. Τώρα σε σχέση με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, δεν το ξέχασα αυτό, αλλά επειδή ανατράπηκε, δεν έγινε προηγουμένως, γιατί πριν να αρχίσουμε τη, συνεδρίαση, η συνάδελφος Λούνατσεκ εξέφρασε τις αντιρρήσεις της σε σχέση με αυτή την ε, αλλαγή άρδιν της ημερήσιας διάταξης και γι' αυτό θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Αρχικά, όταν ε, λάβαμε το προσχέδιο ημερήσιας διάταξης, είχαμε μία συζήτηση για το ε, Αφγανιστάν με τον κύριο Μοριόν και αυτό με έβρισκε σύμφωνη γιατί ήθελα να συζητηθεί. Και μετά ε, απογοητεύτηκα γιατί βγήκε από την ημερήσια διάταξη διότι ο κύριος Μοριόν είναι είτε στο Αφγανιστάν είτε επιστρέφει εδώ. Χαίρομαι που ήμασταν εδώ με τον κύριο Φάιτ και μιλήσαμε για το κοσυφοπέδιο, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από τις άλλες ομάδες και σας κύριε Πρόεδρε και τη Γραμματεία να μας πείτε κατά πόσο η Επίτροπος Φερέρο Βάλτνερ ε, θα μπορέσει να παρευρεθεί αύριο στην Επιτροπή ΑΦΕΤ πριν από την ψηφοφορία για να συζητήσουμε το θέμα της αποστολής αυτής και την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Διαβάσαμε πολλά, ακούσαμε πολλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει τις εκλογές αυτές, στείλαμε παρατηρητές και θα ήταν ιδιαίτερα ε, σκόπιμο και χρήσιμο να έχουμε κάποιον, είτε την κυρία Φερέρο Βάλτνερ, ή κάποιον άλλον από το γραφείο της για μία τουλάχιστον ώρα. Θα ήθελα να με υποστηρίξουν και οι άλλες ομάδες και θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν μπορεί να διοργανωθεί κάτι τέτοιο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σαλαφράνκα, θα ήθελα να διευκρινίσω, κυρία Λούνατσεκ, ότι στην ημερήσια διάταξη Είχαμε την ακρόαση με τον ε, πρέσβη Σέκουι, όχι τον ε, συνάδελφο Μοριών, ο οποίος βρίσκεται in situ για να παρακολουθήσει την διενέργεια των εκλογών και τη λήξη τους. Ο πρεσβευτής Σέκουι είναι υπεύθυνο για θέματα που αφορούν το Αφγανιστάν και το Πακιστάν για να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα σενάρια in loco. Ο πρέσβης δεν είναι εδώ για τον εξής λόγο. Διότι ο Σουηδός Υπουργός Εξωτερικών τον κάλεσε, ο Υπουργός Μπίλτ δηλαδή, και για λόγους ε, σκοπιμότητας ε, παρέμεινε επί τόπου έτσι ώστε να αναπτύξει το, το σενάριο αυτό. Βεβαίως μπορούμε τις επόμενες μέρες να προβλέψουμε κάτι άλλο, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη των πολιτικών ομάδων για να δούμε κατά πόσο μπορεί να συζητηθεί το θέμα με άλλες προσωπικότητες. Ας α, ακούσουμε τη συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ ότι το θέμα είναι ύψης της σημασίας ως προς την εκλογική διαδικασία στο Αφγανιστάν, τη διενέργεια των εκλογών. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε έναν ειδικό αντιπρόσωπο ε, να παρεπερθεί ο ειδικός αντιπρόσωπος στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Ο Φιλίπ Μοριγιόν είναι επικεφαλής της αποστολής των παρατηρητών και ίσως θα μπορούσε να παρεπληθεί εδώ για να μας εξηγήσει την άποψή του. Δυστυχώς, όπως γνωρίζουμε όλοι, γίνεται καταμέτρηση ψήφων και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό αποτελέσμα και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα διενεργηθεί δεύτερος γύρος ή όχι. Με βάση αυτά που ελέγχθησαν και επειδή ο ειδικό αντιπρόσωπος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ στην Επιτροπή μας, με ε, βάση λοιπόν το νήμα της όλης συζήτησης και επειδή αύριο το πρωί θα έχουμε εδώ τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Σχέσεων, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτό το, το θέμα της ε, εκλογικής αναμέτρησης. Βεβαίως είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας και το αφήνω στον πρόεδρο, δηλαδή να κρίνει κατά πόσο μπορεί να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων, δηλαδή να έχουμε παρέμβαση της Επιτρόπου. Θα ξέρουμε πώς έχει γίνει, τι έχει γίνει με την επανακαταμέτρηση και μετά θα μπορέσουμε να αποφανθούμε. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω την θέση του κυρίου Σαλαφράνκα. Αυτό ήθελα. Νομίζω ότι αν ήταν δυνατόν να διευρύνουμε τις συζητήσεις αύριο την ανταλλαγή με τον κύριο Λανταμπούρο για να περιλάβουμε ε, τα θέματα του Αφγανιστάν, νομίζω ότι αυτή θα είναι μια πολύ καλή πρόταση και έτσι δεν θα χάσουμε χρόνο. Διότι ε, δεν είναι πιθανόν, παρόλο που μου αρέσει ε, να έχω ανταλλαγέ με την Επίτροπο Φερεροβάλτερ, αλλά νομίζω ότι μέχρι αύριο δεν θα μπορέσουμε να την έχουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η ιδέα του κυρίου Σαλαφράγκα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Α, με συγχωρείτε. Η κυρία Γκόμες. Απλώς να πω ότι υποστηρίζω και εγώ την πρόταση. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις σας και ε, υποστηρίζω τις προτάσεις σας, όμως για καθαρά οργανωτικούς λόγους ο δόκτωρ Λαντεμπούρου είχε προβλέψει μια συνάντηση ε, μαζί μας για θέματα ενεργειακής ασφάλειας και το θέμα κάθε αυτό ε, είναι άκρο σημαντικό και θα πρέπει να έχουμε, τον, ε, να έχουμε επαρκή χρόνο έτσι ώστε να αναπτυχθεί αύριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια του πρωινού. Εναλλακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τη σκέψη σας, θα πρότεινα να σταθούμε στο θέμα του Αφγανιστάν ή με τον κύριο Λανταμπούρου είτε με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή, με ένα συνεργάτη του δηλαδή. Το απόγευμα μετά την ψηφοφορία. Αυτό δεν θα δημιουργούσε μεγάλες δυσκολίες Νομίζω, ε, αν θέλετε να γίνει αποδεκτή η πρότασή σας και λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας που προβλέπετε το πρωί. Και έτσι, κυρία Λούνα Τσεκ, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είπατε και εσείς και άλλοι, έτσι ώστε να δούμε το κρίσιμο ζήτημα του Αφγανιστάν στην αυριανή μας συνεδρίαση. Δεν ξέρω κατά πόσο ε, ερμηνεύω σωστά αυτά που επιθυμείτε, αλλά έτσι τουλάχιστον κατάλαβα. Ε, η κυρία Λούνατσεκ όμως έχει το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συζητήσουμε αύριο το πρωί το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και να μην συγχαίουμε τα δύο πράγματα, διότι προβλέπουμε ένα δίωρο με τον κύριο Λαντεμπούρου και μετά το θέμα της Μολδαβίας. Γι' αυτό συμφωνώ με αυτά που είπε ο πρόεδρός μας, δηλαδή να γίνει συζήτηση το απόγευμα. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να παρευρεθεί εδώ η κυρία Φέρερο Βάλτνερ. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά θα ήθελα να ε, σας ζητήσω να το προσπαθήσετε. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθεί η γραμματεία. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Πρόεδρος, δεχόμαστε αυτή την πρόταση σαν πρόταση και θα ορίσουμε την αυριανή ημερήσια διάταξη με αυτές τις ε, επιθυμίες όπως διαμορφώθηκαν. Ας περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, τμήμα 3 του προϋπολογισμού 2010 Επιτροπή χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή. Σας ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Νέιτς, στη συντάκτρια γνωμοδότησης. Και μετά θα παρέμβουν οι βουλευτές. Έχει το λόγο η συντάκτρια. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα κάνω παρατηρήσεις πάνω στο γεγονός ότι υπάρχουν τώρα λιγότεροι συνάδελφοι για τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό από ότι είχαμε για την ουσία της πολιτικής απλώς. Θα ήθελα να τονίσω ότι χωρίς οικονομικά μέσα δεν μπορεί κανείς να έχει καμιά πολιτική. Αλλά αυτά ως εισαγωγή. Πρώτη παρατήρηση σχετικά με την στήλη 4 που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, συνομιλητής, ως εταίρος παγκόσμιος. Θα ήθελα να πω ότι τα σχέδια αυτά έχουν πολύ λίγη χρηματοδότηση και αυτή είναι η περίπτωση εδώ και μερικά χρόνια. Έχουμε όμως ε, μερικούς λόγους ικανοποίησης, διότι αυτό που προβλέπεται στην περίπτωση των περιφερειακών προϋπολογισμών θα πρέπει να το ενισχύσουμε στην Ευρώπη κυρίως όσον αφορά την βοήθεια στην προενταξιακή περίοδο για την μεταφορά, την ενέργεια, την ε, παιδεία, τα μέτρα συμφιλίωσης και για την πρόθεση της αηφόρου οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Εξακολουθούμε ε, να εκφράζουμε την υποστήριξή μας αν συμφωνείτε ούτως ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία ενδελεχή που θα βασίζεται σε δύο πυλώνες, δηλαδή τις εταιρικέ σχέσεις, τις ανατολικές και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Αλλά και εδώ επίσης φοβούμεθα ότι οι πιστώσεις που προβλέπονται δεν θα είναι επαρκείς. Εκτός από αυτά, ζητούμε μια στρατηγική σαφέστατη όσον αφορά στην Παλαιστίνη όπου η οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνοδεύεται με έναν ισχυμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Τονίζουμε επίσης ότι η μείωση της ε, οικονομικής βοήθειας στην Παλαιστίνη δεν θα ήταν κάτι το ρεαλιστικό και δεν θα αντανακλούσε την πολιτική σημασία που έχει η Μέση Ανατολή για μας. Ζητούμε λοιπόν από την Κομισιό να μην αργήσει να παρουσιάσει τις προτάσεις σχετικά με τις δαπάνες που απορρέουν από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το Μάρτιο 2009 στην διάσκεψη των δωρητών του Σάρμελ Σέχ. Οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν. Θα θέλαμε επίση να υπενθυμίσουμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ότι το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι για μα μια πολιτική προτεραιότητα απόλυτη και λυπούμεθα άλλη μια φορά για τι περικοπές που προτείνονται. Επισύρουμε την προσοχή του Συμβουλίου και τη Κομισιόν πάνω στις διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα της Κύπρου. Για την ώρα οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν φαίνεται ότι προοδεύουν καλά, ότι εξελίσσονται ικανοποιητικά. Νομίζουμε ότι η βοήθεια στην τουρκική κοινότητα πρέπει να συνεχιστεί. Για να κλείσω, Πιστεύω προσωπικά, ελπίζω μάλλον, ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα επικυρωθεί και θα τεθεί σε ισχύ. Αν αυτό γίνει, αυτό θα έχει συνέπειες σημαντικές για την εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική ασφαλείας και αυτό θα επισύρει συμπληρωματικές δαπάνες που για την ώρα δεν έχουν προβλεφθεί. Για να κλείσω, θα ήθελα άλλη μια φορά να τονίσω ότι ότι οι πιστώσεις ε, οι οποίες είναι ανεπαρκείς ε, για τον τίτλο 4 μπορεί να αποτελέσουν ε, αντικείμενο πιέσεων εάν υπάρξουν άλλες θεσμικές τροποποιήσεις και νομίζω ότι αν η συνθήκη τεθεί σε ισχύ θα πρέπει να εξαγάγουμε τις οικονομικές συνέπειες αμέσως όταν γίνει η αξιολόγηση των δημοσιονομικών προπτικών. Επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι ζητούμε από την Κομισιό να μην χρησιμοποιήσει το αποθεματικό της κατεπίγουσας βοήθειας για δραστηριότητες μακροπρόθεσμες και εδώ είμαστε απογοητευμένοι διότι στον τίτλο 4 προβλέπεται πολύ μικρό περιθώριο. Όλα αυτά μου φαίνονται ουτοπικά. Αν έχει κανείς ένα μικρό περιθώριο, τίποτα από τα προβλεπόμενα δεν θα γίνουν, αλλά δεν λειτουργούν τα πράγματα έτσι. Κάθε φορά έχουμε απρόβλεπτα γεγονότα. Θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά να κάνουμε ακροβασίες δημοσιονομικές, αν θέλουμε να έχουμε τα απαιτούμενα δημοσιονομικά μέσα. Φοβούμαστε ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός για το 2010. Οι περισσότερες τροπολογίες τις οποίες προτείνω έχουν ως στόχο να αμφιζ να θέσουν ένα αμφιβόλο της τροποποίησης που προτάθηκαν. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω σε μια τροπολογία συμβιβαστική για το 190604. Αν υπάρξει μια νέα διατύπωση αυτής της γραμμής, θα μπορούσα να δεχθώ αυτό το, την πρόταση για να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο Ινστιτούτων Εκπαίδευσης ε, για την διαχείριση ε, των πολιτικών κρίσεων όσον αφορά τις ειρηνευτικές αποστολές ε, και την διευθέτηση των κρίσεων μετά από συγκρούσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Νέιτς για την παρουσίασή και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια. Η ομάδα μου υποστηρίζει τη γενική γραμμή της εισηγήτριας και είμαι ένας από εκείνους που έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία από το θέμα. Είναι ε, ε, μια πειρά 11 ετών. Δύο σημεία μπορούν να αναφερθούν. Υποχρηματοδότηση κατηγορίας 4, δεν έχει αλλάξει αυτή. Και κάθε χρόνο ένα δεύτερο σημείο που το λέμε πάντα με κριτικό πνεύμα είναι το γελίο ποσό της χρηματοδότησης ε, στην Παλαιστίνη. Κάθε χρόνο το βλέπουμε. Ε, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δίνουμε τα διπλάσια και πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε από πού θα τα πάρουμε τα κονδύλια. Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε πιο ρεαλιστές στα ποσά που αναγράφουμε. Ε, τα λέμε και τα ξαναλέμε και πάντοτε βγαίνουμε αληθινοί. Αλλά φαίνεται ότι δεν μας ακούει κανείς. Τέλος πάντων, στα πλαίσια του ψηφίσματος ε, θα ήθελα να πω Δεν συμφωνούμε με την τροπολογία 4 που υποστηρίζει η συγγήτρια, γιατί ναι με το gender mainstreaming το βλέπουμε ως σημαντική πολιτική δραστηριότητα, αλλά το σημείο κλειδί των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι, ε, μην, ε, είναι λίγο υπερτιμημένο. Δεν είμαστε λοιπόν υπέρ της ε, τροπολογίας 4. Τώρα, η τροπολογία Van Orden. διευκρινίζει κάπως περισσότερο το θέμα των Τουρκοκυπρίων και των πιστώσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί προς τα εκεί. Είναι μια υπόδειξη. Ο συνάδελφος Κασουλίδης μου φώναξε ότι μέχρι τώρα ήταν στη φάση του σχεδιασμού και τώρα καταβάλλονται ουσιαστικά, κανονικά τα χρήματα, το λαμβάνω υπόψη μου αυτό, αλλά θα ήθελα να πάει λίγο πιο γρήγορα αυτό το πράγμα και να φτάσουν τα χρήματα εκεί στους αποδέκτες που τα χρειάζονται. Αυτά για το ψήφισμα. Τώρα, για τις τροπολογίες για τον προϋπολογισμό συμφωνούμε με τη γραμμή πλεύσης της εισηγήτριας σε μεγάλο βαθμό με τις πολιτικές προτεραιότητες στην πολιτική γειτονία και τη Μέση Ανατολή, την Εγγύς Ανατολή. Ε, βεβαίως υπάρχουν και άλλα βασικά θέματα που πρέπει να κάνουμε στον κόσμο, αλλά αυτά είναι οι δύο προτεραιότητες που πρέπει να αναδειχθούν. Ε, επίσης είμαστε και εμείς υπέρ του να υποστηριχθεί το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν, τα ποσά που αναγράφει. Ε, το, έργο το, το είναι μια, ένα παιχνίδι που παίζεται κάθε χρονιά με το Συμβούλιο, που κατεβάζει τα ποσά, τα μειώνει, πρέπει να τα ξαναβάλουμε. Ε, τώρα, αντίθετα με την εισηγήτρια, πιστεύουμε ότι πρέπει ως εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ειδικό εκπρόσωπος να είναι ο πλέον, η πλέον ενδεδειγμένη προσωπικότητα. Αυτό είναι ε, σημαντικό να φτάσουμε ε, να τον επιλέξουμε, αλλά θα πρέπει να είναι το καλύτερο, το πλέον ενδεδειγμένο πρόσωπο πέρα από το φύλλο. Επίσης, το Senior Expert Service που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ε, νότερα ειδικά στελέχη, εμπειρογνώμονες, οι ανώτεροι εμπειρογνώμονε και ω εταίροι σε προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την Κομισιόν και να συμμετέχουν, γιατί σε αυτά τα θέματα χρειάζεται μεγάλη εμπειρία ε, και θα πρέπει αυτή να ε, διοχετεύεται και στα επιμέρους προγράμματα στα οποία θα ενταχθούν οι ειδικοί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράγκα έχει στη συνέχεια το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία ε, Νέης για την εξαιρετική εργασία κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πρόκειται για μία δύσκολη διαδικασία μέσα στα πλαίσια της αλλαγής αυτής της ε, θητείας και γι' αυτό υπήρχαν και επιπρόσθετες δυσκολίες. Ο κύριος Γκάλερ ε, μίλησε πολύ σωστά για τη θέση της ομάδας μας. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν διάφορες προτεραιότητες και ε, εναλλαγές, εναλλακτικές λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις εναλλακτικές που προβάλλονται και υπάρχει ένα σημείο επί το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γκάλερ, δηλαδή την ε, δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με εμπειρογνώμονες, με τους ε, seniors, και αυτοί οι seniors θα μπορούσαν να μας ε, διαθέσουν τη γνώση τους πάντα η ΑΦΕΤ και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε υποστηρίξει αυτή την τάση διότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό αντίκρισμα και θα μπορούσαμε να δείξουμε την καλή μας θέληση σε σχέση με την τροπολογία 55 για το μέσο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς δεχόμαστε τις προσπάθειες του κυρίου Γκάλερ, άρα θα αποσύρω το πρώτο τμήμα της τροπολογίας μας, της τροπολογίας μου, για να διευκολύνω μια συνεννόηση. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε με την πρόταση της εισηγήτριας και την πρόταση του κυρίου Γκάλερ. Ευχαριστούμε κύριε Σαλαφράκα. Ο κύριος Λέζινγκ έχει το λόγο. Η κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την προσεκτική δουλειά που μας έκανε. Πολλές φορές λέμε ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν επαρκούν για να γίνουν σοβαρές ε, Δουλειέ στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Σε αυτά τα πλαίσια αναφέρομαι στην παρέμβασή μου στην τελευταία συνεδρίαση της ΑΦΕΤ, όπου ετώνησα ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστώσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, στα πλαίσια στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράδειγμα το πρόγραμμα Γαλιλαίο από τον προϋπολογισμό το γεωργικό αναφέρθηκε ότι στο μέλλον ενδεχομένως μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας θα δίνονται περισσότερα λεφτά για τους εξοπλισμούς. Αναφέρθηκε ότι υπάρχει ελπίδα να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό και επειδή μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης θα ε, αυξάνονται οι εξοπλισμοί, εμείς απορρίπτουμε τη συνθήκη αυτή ως ε, παράταξη. Τα χρήματα αυτά τα χρειαζόμαστε για πολλούς άλλους τομείς και εξακολουθούμε να θέλουμε μείωση των εξοπλισμών υπέρ των κοινωνικών έργων. Και σήμερα θέλουμε να σταματήσει η παράνομη χρήση κοινοτικών κονδυλίων για προγράμματα ε, στρατιωτικής φύσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Η κυρία Χαπταλά έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Νέιτς επέμεινε επί του γεγονότος ότι όλες αυτές οι εξωτερικές δραστηριότητες υποχρηματοδοτούνται. Εργάστηκε εξαίρετα και αυτό το λέω ε, εξ ονόματος ολόκληρης της ομάδας των Πρασίνων. Σε σχέση με αυτό το σχέδιο ψηφοφορίας ε, υπάρχει τροπολογία 4 η οποία αναφέρθηκε. Μιλάμε για το γεγονός ότι σύμφωνα με την ε, Ευρωπαϊκή Συνθήκη θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Μιλάμε για mainstreaming για όλες τις εξωτερικές πολιτικές. Άρα αυτή η τροπολογία μου φαίνεται εξαιρετική. Τώρα, ως προς τις άλλες ε, προτάσεις, ε, δημοσιονομικές προτάσεις, καταρχήν να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, διότι έλαβε υπόψη τις μη κυβερνητικές και τα πιλωτικά σχέδια. υπάρχει ένα μέσο χρηματοδότηση στα πλαίσια των εξωτερικών υποθέσεων που επέτρεψε αυτή τη δράση των μη κυβερνητικών. Είναι το μέσο σταθερότητας. Θεωρώ ότι η εισηγήτριά μας βλέπει θετικά αυτά που προτείναμε εμείς ως πράσινοι για τον Κάφκασο. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα πιο, αυτές είναι οι πιο σημαντικές τροπολογίες που μας απασχόλησαν. Ευχαριστούμε την κυρία Χάουταλα. Μάντλενερ. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου σας παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μιλάω εξ ονόματος μιας ομάδας, αλλά εξ ονόματος του δεύτερου κόμματος ε, στις κάτω χώρες ε, στις ευρωεκλογές. Ε, για μας ε, το προϋπολογισμός είναι θέμα κρατών και όχι κοινοβουλίου. Οι διπάνες αυξάνονται. Ποιος θα πληρώσει ε, την, το λογαριασμό, οι φορολογούμενοι των ευρωπαϊκών χωρών που, ε, είναι, που συνεισφέρουν περισσότερο. που, και όπως ξέρετε οι κάτω χώρες συνεισφέρουν περισσότερο και θέλω να διαμαρτυρηθώ. Απογοητευόμεθα από τα χρήματα που στέλνονται στην Παλαιστίνη πρόκειται για ένα κονδύλια τελείωτα για μας. Δεν θα έπρεπε να δώσουμε στα εδάφη της Παλαιστίνης ούτε ένα ευρώ. Θα ψηφίσουμε κατά του ψηφίσματος αυτού και ζητώ από όλου να κάνουν το ίδιο. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μάντλερ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης εισηγητής της ομάδας μας δεν μπόρεσε να είναι εδώ, πάντως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μέσα στην ομάδα μας. Συμφωνώ με την προσέγγιση της εισηγήτριας. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες για την εκπόνηση αυτής της γνωμοδότησης. Μερικές παρατηρήσεις τώρα. Δυστυχώς είμαστε απογοητευμένοι διότι το ΕΛΚ δεν μπορεί να υιοθετήσει την τροπολογία 4 σχετικά με την ισότητα μεταξύ φύλων, όπου είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο εξωτερική πολιτική, αφορά όλες τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λοιπά ή της ανάπτυξης. Άλλη παρατήρηση, η στρατηγική στη Βαλτική Έχουμε μερικές αμφιβολίες ως προς τον εξωτερικό χαρακτήρα της Βαλτικής. Είναι μάλλον εσωτερική πολιτική η Βαλτική, έτσι δεν είναι, σχετικά ε, με το πιλωτικό σχέδιο των Πρασίνων, σχετικά με την, τον εκδημοκρατισμό. Καταρχήν συμφωνούμε, συμφωνούμε για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, αλλά Νομίζω ότι αυτό είναι κατακαιρματισμός σε πολλές γραμμές του προϋπολογισμού. Είναι μια κονιορτοποίηση. Ε, ε υπάρχουν επίσης άλλες παρατηρήσεις, παρατηρήσεις του ΕΛΚΑ για τις ε, τροπολογίες. Έχουμε μια αναφορά στην Κούβα, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πρόοδοι προς τον εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα. Αλλά νομίζω ότι στις παρατηρήσεις αυτές ε, δεν αναφέρω καμιά χώρα. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον εκδημοκρατισμό ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά εάν αναφέρουμε μια χώρα συγκεκριμένα, αυτό δημιουργεί προβλήματα. Και αυτό μπορεί να έχει αρνητική εξέλιξη για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πάντως την εισηγήτρια για την πρότασή σας. Ευχαριστώ. Κυρία Μίνιτς. Ο κύριος Βαν Όρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο καλός συνάδελφος από τις κατοχώρες είπε ότι ε, είναι ε, καθαροί συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό και εμείς. Νομίζω ότι πρώτα είναι η Γερμανία, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και τρίτος ε, νομίζω συνεισφέρον είναι οι κατοχώρες. Βεβαίως ε, αυξάνεται ε, η συνεισφορά του Ηνωμένου ε, Βασιλείου μετά τον κύριο Μπλερ. Αλλά αφήνω αυτές τις παρατηρήσεις κατά μέρος. Πολύ καλά. Ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση. Κύριε Βαν Όρντεν, μαθηματική διευκρίνηση. Κυρία εισηγήτρια, σας ξαναδίνω τον λόγο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να λάβει το λόγο από πλευράς της Κομισιό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ που με συγχαρήκατε για αυτή την εργασία και εγώ ευχαριστώ την γραμματεία της Επιτροπής η οποία συνέβαλε σημαντικά στο έργο αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις είπατε ότι είσαστε υπέρ των μεγάλων γραμμών της εκθεσής μου. Αύριο το πρωί θα προσπαθήσω να συζητήσω με τον κύριο Σαλαφράνκα για την τροπολογία 50-51. Να επανέλθουμε στο θέμα αυτό ε, ε, των δικτύων των σενιόρ. Ίσως τα πράγματα δεν είναι πολύ σαφή. Πρέπει να πω ότι εκπλήσωμε διότι ο κύριος Γκαλά μας είπε ότι ε, το ΕΛΚ ψήφισε κατά της τροπολογίας 4. Ίσως πάει λίγο μακριά το πράγμα. Αλλά έχουμε 12 εκπροσώπους ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα. Πιστεύω ότι ίσως μόνο αρμόδιοι είναι οι άνδρες και δεν υπάρχει καμία γυναίκα που να είναι αρκετά αρμόδια ε, για μία από αυτές τις θέσεις. Σας ζητώ άλλη μια φορά να σκεφτείτε το θέμα αυτό. Δεν θέλω να επανέλθω στη συζήτηση για να δούμε αν μια χώρα είναι καθαρό συνεισφέρον ή όχι. Αυτή η συζήτηση δεν θα είχε κανένα τέλος, θα ήταν ατελείωτη. Ε, έχουμε στις διάφορες γλώσσες μας διάφορες εκφράσεις. Υπάρχει η γαλλική αριθμητική, ο τρόπος ο ολλανδικός υπολογισμού. Όλες αυτές οι εκφράσεις έχουν ως συνέπεια ο καθένας ε, να ευνοεί τον εαυτό του, να ε, μιλάει για τον εαυτό του ανάλογα με τις ανάγκες της χώρας. Το αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ευρωπαϊκό. Αν χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το επιχείρημα, πότε δεν θα τελειώσουμε στη συζήτησή μας. Θα συζητήσω και με τον κύριο Σαλαφράνκα και πάλι ευχαριστώ τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και θα ήθελα... Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε χωρίς δυστολία να υιοθετήσουμε τις διάφορες τροπολογίες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και όσους έλαβαν το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Όπως ξέρετε θα ψηφίσουμε αύριο το απόγευμα σχετικά με τη γνωμοδότηση αυτή. Τώρα θα ασχοληθούμε με τα σημεία 7 και 8, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με το Τατζικιστάν πρόταση ψηφίσματος και συμφωνία εταιρική σχέσης. Υπάρχουν μερικές τροπολογίες που θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Για τα δύο αυτά σημεία ο κύριος Πέτερ είναι ο εισηγητής και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Φαίνεται ότι πλησιάζομαι στην ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Δεν θα επαναλάβω όλους τους λόγους για τους οποίες πρέπει να είμαστε υπέρ αυτής της ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Την περιμέναμε εδώ και καιρό, ότι άλλαξε από τον Ιούλιο και μετά. Τα κράτη-μέλη ολοκλήρωσαν τις ε, διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο και τώρα ήρθε η ώρα να συγκατατεθεί και το Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχουν 57 ε, τροπολογίες συνολικά που νομίζω ότι παραμπαίνουν σε λεπτομέρειες, ε, το κάνουν πολύ επακριβές στο κείμενο, άλλες τροπολογίες αναφέρονται στις εξελίξεις των τελευταίων ε, μηνών, κάποιες άλλες είναι λίγο υπερβολικές και δεν έχουν και τόση σημασία αφού δεν είναι σχετικές, δεν αναφέρονται στη συγκεκριμένη συμφωνία θέλουν μέσω της συμφωνίας να προωθήσουν ε, άλλου είδους συμφωνίες. Ε, εγώ έχω εγκρίνει τις περισσότερες τροπολογίες που είναι σχετικές. Ε, ευχαριστώ την Κομισιόν, συνεργάστηκα πολύ καλά μαζί της και επίσης ευχαριστώ την πρεσβεία του Τατζίκισταν γιατί και με την πρεσβεία έκανα πολλές χρήσιμες συζητήσεις. Θα μπορούσα να μπω και να σχολιάσω κάθε μία τροπολογία χωριστά αλλά ε, επειδή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, ε, δεν νομίζω να υπάρχει ανάγκη. Ο, ε, ναι. Οι τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στην χρήση των πόρων, των υδάτινων πόρων, έχουν περιληφθεί στις τροπολογίες 29 και 30 και σε σχέση με τα βασανιστήρια αναφέρονται στις τροπολογίες 50 και 51. Η τροπολογία 38 είναι μια τροπολογία η οποία θα μπορούσε να αλλάξει διότι πρόκειται για το θέμα του ελέγχου των ε, χρηματοοικονομικών, ε, της χρηματοοικονομικής αρρωγής. Οι πράσινοι προτείνουν, ε, προτείνουν έναν λεπτομεριακό καταμερισμό αυτού του θέματος, αλλά δέχουμε και τη θέση της Επιτροπής που θεωρεί ότι δεν χρειάζεται να εισαγάγουμε νέα μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πούν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την τροπολογία 53 Λαντσπέργης. Εδώ μπορώ να πω ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, άρα ε, δεν χρειάζεται, είναι περιττή αυτή η τροπολογία. Ευχαριστούμε τον κύριο Πέτερλε. Το λόγο έχει η κυρία Κοπά. Μια Κύριε συνάδελφοι, κανεί από εμά δεν μπορεί να υποστηρίξει πιστικά ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία στο Τατζικιστάν είναι ικανοποιητική. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο, μέσα από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να γίνεται απόλυτα σαφέ ότι η συγκατάθεση και αποδοχή τη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία αποτελεί πάνω απ' όλα μια κίνηση καλή θέληση από μέρους μας και πως η ενισχυμένη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει ουσιαστική βελτίωση σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Πιστεύω πως το μήνυμα αυτό υπάρχει στο ψήφισμα που ετοίμασε ο συνάδελφος Πέτριλε και θέλω να τον ευχαριστήσω για τη δουλειά του. Με δύο τροπολογίες που κατέθεσα, επέλεξα να θέσω ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, που είναι η συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Η υποχρέωση για συνεργασία αναφέρεται στο άρθρο 70 της εταιρικής σχέσης με το Τατζικιστάν, όμως στην πρόταση ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας δεν γίνεται καμία αναφορά στην πολιτική μας στον τομέα αυτό. Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί πως το κείμενο της εταιρικής σχέσης δεν ρυθμίζει λεπτομερώς το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και της επανεισδοχής, αλλά ζητάει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ξεχωριστή ειδική συμφωνίας. Θεωρώ πω πρέπει να το τονίσουμε αυτό στην έκθεσή μα και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να προωθήσει τι σχετικέ διεργασίες, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί κηρύτρα επανεισδοχή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθιστε να συμπεριλαμβάνει σε παρόμοιε συμφωνίε με τρίτε χώρε. Πρέπει με άλλα λόγια να επανέλθουμε, και αυτό γενικότερα και όχι μόνο στην περίπτωση του Τατζικιστάν, στι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη Σεβίλη που ήδη από το 2002 ζήτησε να τίθεται ως προϋπόθεση για τη σύσφυξη στενότερων σχέσεων με τρίτες χώρες το ζήτημα της κοινή διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και της υποχρεωτικής επαναπροώθησης σε περίπτωση παράνομης μετανάστευσης, πάντα φυσικά με σεβασμό για τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κοπά. Λέζιν. Μια φακολτά. Ja, ich kann gleich an die Ausführung Συνεχίζω και που σταμάτησε η προηγούμενη συνάδελφος. Ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε για την πολύ διεξοδική έκθεση. Η ομάδα μου, Γκουε, ε, έχει προβλήματα με την εταιρική σχέση που δεν μπορούν εύκολα να επιληθούν με τις προτάσεις που γίνονται και με τις τροπολογίες. Γιατί οι τομείς που μας ενδιαφέρουν δεν αναφέρονται καθόλου σε αυτό το πρόγραμμα, ε, στο σχέδιο σύστασης. Όμως ε, αναφέρθηκε ότι σε κάθε εταιρική σχέση υπάρχει ένα δούνε και λαβίν και από τις δύο πλευρές. Αλλά αναρωτιέμαι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, λαμβάνονται υπόψη. Ε, καταρχήν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα μακρά σύνορα Τατζικιστάν, Αφγανιστάν, την διεύρυνση του πολέμου που απειλεί να γίνει ένας νέος πόλεμος του Βιετνάμ, ε, ο τεράστιος αριθμός προσφύγων. Στην Ουκρανία το, η διεθνής διαχείριση των προβλημάτων ε, προσφύγων θα συμπεριλάβει και το Τατζικιστάν. Ε, θα, υπάρξουν, θα υπάρξει δημιουργία καταβλισμών προσφύγων στο Τατζικιστάν για να λάβει υπόψη τα ρεύματα των, τις ροές των προσφύγων. Επίσης, ε, αναρωτιόμαστε σε σχέση με τη Συμφωνία εταιρική Σχέσης υπάρχει ε, και μια ειδικότερη πρόβλεψη που θα αφορά τους στο καθεστώς και την αντιμετώπιση των προσφύγων. Ε, το 2007 είχαμε κάνει κάτι παρόμοιο με την Ουκρανία. Όπως είπε και η συνάδελφος προηγουμένως, ε, μια συμφωνία επανεισδοχής ε, των ε, μεταναστών, μεταναστριών προβλέπεται. Αναφέρθηκα στα μακρά σύνορα, 1200 χιλιόμετρα σύνορα με το Αφγανιστάν. Στην πρόταση ψηφίσματος λέει ότι λόγω των σύνορων αυτών το Τατζικιστάν αποκτά στρατηγική σημασία. Και αναρωτιόμαστε το Τατζικιστάν συγκεκριμένα τι ρόλο θα παίξει σε σχέση με τον πόλεμο του Αφγανιστάν θα διαθέσει βάσεις για τα στρατεύματα των δυτικών, θα είναι χώρα διέλευσης των ε, δυτικών στρατευμάτων, ε, θα δράσει ο, η κατάσταση στο Αφγανιστάν αποσταθεροποιητικά στο Τατζικιστάν. Τέλος, μια ερώτηση που, αφορά την οικονομία. Η, η συμφωνία εταιριστική σχέση μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών όπως το Τατζικιστάν ε, αποσκοπούν στη δημιουργία ζώνης συναλλαγών. Ε, για να βελτιωθεί και η θέση των δυτικών επιχειρήσεων. Αναρωτιόμαστε πάνω σε αυτή τη βάση πώς ε, πρέπει να καταλάβουμε το, αυτό που λέει ότι θα πρέπει να γίνουν διαθροτικές αλλαγές στο Τατζικιστάν για την προώθηση των ξένων επενδύσεων. Τι μέτρα δηλαδή συγκεκριμένα έχουν υπόψη τους. Υπάρχουν ήδη κάποιες πρόοδοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι βήματα κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αν δεν απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, δεν μπορούμε να κρίνουμε τη συμφωνία. Ούτε μπορούμε να συμφωνήσουμε με την πρόταση ψηφίσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λόζινγκ. Η κυρία Χάουταλα έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Είμαι ικανοποιημένη με τον τρόπο που ο εισηγητής αντιμετώπισε το θέμα και πώς αντιμετώπισε και επίσης τις τροπολογίες των πρασίνων. Πρότεινε συμβιβασμό στο συμβιβασμό 1 και 2 που μας φαίνονται εξαίρετοι. Μένει ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με το 8α της κυρίας Λόζινγκ τι εννοούμε στα πλαίσια του Τσατατζικιστάν όταν μιλάμε για δομές. Μετά έχετε άλλες τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν από τους πράσινους σχετικά με τις δημοσιονομικές βοήθειες και τις άλλες βοήθειες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με καλό τρόπο. Μιλάμε για μια ομάδα παρακολούθησης. Ε, τι, τι είναι αυτό. Ε, μπορείτε ε, να μας πείτε περί τίνος πρόκειται, διότι οι δωρητές θέλουν να ξέρουν ποια είναι τα κριτήρια για να χρησιμοποιηθούν με καλό τρόπο αυτές οι ενισχύσεις. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την ομάδα παρακολούθησης. Νομίζω ότι πρόκειται για την ε, τροπολογία 38. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα. Επειδή ζητήθηκαν ε, απαντήσει από την Επιτροπή, ο δόκτωρ Μπέρν έχει το λόγο για να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ε, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε ήδη πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να τα καλύψω όλα στο χρόνο που έχουμε. Καταρχήν είμαι ευγνώμων στον κύριο Πέτερλε για την πολύ εμπεριστατωμένη στέρεη δουλειά στα πλαίσια του ψηφίσματος και της τροπολογίας ορισμένες εκ των οποίων πρέπει να σχολιαστούν. Αρχίζω με την 38 που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ίσως δεν βλέπουν όλοι ότι αυτό που λέει είναι ότι δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο μεταξύ, ε, από την Κομισιόν για την παροχή βοήθειας στο Τζικιστάν με τις ε, ε, κυρώσεις και, τις, ε, ε, και τα κίνητρα. Εκπλήσω με αυτό που λέει, γιατί η Κομισιόν κατανοεί βέβαια την πρόθεση της τροπολογίας, αλλά χρειάζεται βεβαίως συνεννόηση μεταξύ όλων των δωρητών για κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε ότι η υφιστάμενη συνεργασία που έχουμε με τους διεθνείς δωρητές που περιλαμβάνει την Παγκόσμια Τράπεζα, τη, τα Ηνωμένα Έθνη κλπ. που έχουμε συμφωνίες μαζί τους και εκεί κινούμεθα, δίνει καλή, καλές προϋποθέσεις για συνεργασία και επίσης ε, έχουμε και την ομάδα στήριξης ε, που περιλαμβάνει όλους τους διεθνείς δωρητές και που συναντιέται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ε, οι δωρητές με τους οποίους συνεργάζεται η Κομισιόν. Εμείς ε, ε, τώρα έχουμε το, το νέο κανονισμό DCI και τους θεματικούς προϋπολογισμούς, συνεργασία τάσης που την λαμβάνουμε υπόψη και έτσι έχουμε τη νομική βάση για τη συνεργασία μας για την Κεντρική Ασία. Σε ό,τι αφορά τώρα την παρακολούθηση, αυτό που προτείνεται από την Κομισιόν είναι οι ευρωπαϊκές προσφορές ε, ε, να αξιολογούνται από μια ειδική μονάδα που μαζί με την αντιπροσωπεία στο επιτόπου ε, θα συνεργάζονται αποτελεσματικά. Μπορεί να δημιουργηθούν κάποιε δυσκολίε γιατί το υφιστάμενο πλαίσιο συνεργασία, το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε, ε, μα φτάνει για να ανταποκριθούμε στις ε, ευθύνες και αρμοδιότητές μας στο, και στο Τατζικιστάν ειδικότερα και στην Κεντρική Ασία γενικότερα. Τώρα κάποιες άλλες παρατηρήσεις που έγιναν. και αυτά που είπε η κυρία Κοπά, ε, το PCA και το παράνομο εμπόριο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται ο ΑΣΕ και διάβασα σήμερα μάλιστα ότι έγιναν επισκέψεις στην Ευρώπη και στη Βιέννη στους αρμόδιους οργανισμούς Πολλά από αυτά τα θέματα όμως που αφορούν την παράνομη μετανάστευση αναπτύχθηκαν στα πλαίσια μιας κατάστασης μετά το PCA, τη ε, εταιρική σχέση. Ε, η Κομισιόν δούλεψε πάνω σε πιο περιορισμένη βάση ευθύνης ε, σε σχέση με το πόσο μακριά μπορούμε να πάμε. Αν υποθέσουμε ότι θα υπάρξει νέα συμφωνία PCA, μπορεί να προβλέψει βαθύτερη συνεργασία σε μεγαλύτερο βάθος, ευρύτερη. Θα υπάρξουν κοινέ επιτροπές για την ε, οικονομική συνεργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα θέματα. Και επίσης Πολλές από τις ανησυχίες που εκφράζονται από τα, μέσα από τα σχόλια αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να ειδωθούν καλύτερα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επανεισδοχής που οπωσδήποτε θα συζητηθεί μετά την υιοθέτηση των συμφωνιών PCA, εταιρική σχέση και συνεργασία. Θα συζητηθούν λεπτομερέστερα και θα υπάρξουν και διαβουλεύσεις με τους οργανισμούς όπως Frontex κλπ. Ε, εκεί είναι το κατάλληλο πλαίσιο. Το άλλο θέμα που έθεσε η κυρία Λέζινγκ, δηλαδή ροές προσφύγων, Υπάρχει μια ανησυχία προφανώς και ο ρόλος του Τατζικιστάν και με το γιατί ο πρόεδρος Μπαρόζο επισκέφθηκε τον πρόεδρο του Τατζικιστάν και είπε ο πρόεδρος του Τατζικιστάν ότι θεωρεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ε, περιφερειακή ασφάλεια και συνεργασία και θεωρεί ότι είναι, αν θέλετε, μια ουδέτερη, ένα ουδέτερο κράτος ε, που θα αντισταθεί στην τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό, την ε, το παράνομο εμπόριο και έτσι μπαίνουμε σε, στην ουσία της συνεργασίας με το Τζικιστάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την διασυνοριακή ασφάλεια και οπωσδήποτε θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, αυτό το κάνουμε ε, με, το, με ένα πρόγραμμα που άρχισε το 2001 ε, στο Τζικιστάν και απεδείχθη πολύ αποτελεσματικό και σήμερα το απόγευμα μάλιστα υπάρχει μια συνάντηση για το Αφγανιστάν όπου εκπρόσωπος της UNDP μιλούσε για το ε, Bomb Buffer Agreement το οποίο είναι το αντίστοιχο για να ε, φροντίσει για την ασφάλεια από την πλευρά του Αφγανιστάν. Θέλουμε λοιπόν καλύτερη συνεργασία και μεταξύ των δύο χωρών για καλύτερη αντιμετώπιση της ασφάλειας των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, αυτό οπωσδήποτε ε, ενδιαφέρει στα πλαίσια ενός σεναρίου μετά την ε, Συμφωνία PCA. Η Κομισιόν θέλει να αναπτυχθεί ο ιδιωτικό τομέα είναι τομέας εστίασης ε, συγκεκριμένη στην περίοδο 2007-2013. Ήδη η Κομισιόν ε, παρέσχει υποστήριξη ε, στον ιδιωτικό τομέα για να δημιουργηθούν μονοθυριδικές υπηρεσίες και να μπορούν να διευκολύνουν οι ξένοι επενδυτές να παίρνουν τις πληροφορίες που θέλουν για να επενδύσουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, στα πλαίσια του οικονομικού κλίματος που προωθούμε στο Τατζικιστάν και το οποίο επηρεάστηκε ε, δυσμενώς από την μείωση των εμβασμάτων από τη Ρωσία. Υπάρχει μείωση 40% ε, κάθε χρόνο και αυτό επηρεάζει δυσμενέστατα την ικανότητα της κυβέρνησης του Τατζικιστάν να ανταποκριθεί στις ευθύνες της στον τομέα της υγείας, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής και μάλιστα έχουμε ε, αιτήσει ε, για παροχή 30 εκατομμυρίων. Αυτό το αίτημα υπευλήθη στον Επίτροπο Αλμούνια. Μακάρι να ε, τύχει θετικής αντιμετώπισης από την Κομισιόν και τους Επιτρόπους. Αυτά είναι τα βασικά. Ελπίζω να μην παρέλειψα τίποτε. Ζητώ συγγνώμη αν παρέλειψα και ευχαρίστω να απαντήσω και στις πληρωματικές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δόκτωρα Μπέρν για τα τελικά σχόλια. Ο κύριος Πέτερ έχει το λόγο, ο εισηγητής. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν, καθώς και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διασαφήσεις αυτές. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες ε, των συνοδέλφων σε σχέση με αυτά τα επιμέρους ε, θέματα σκοπιμότητας. Μιλάμε για τις ε, δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της συμφωνίας. Δηλαδή μιλάμε για την αρχή αυτής της συμφωνίας υπάρχει μία ρήτρα διασφάλισης η οποία θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Άρα δεν πρέπει να επιβαρύνουμε αυτή την έκθεση με, περισσότερα, με, περισσότερο κείμενο, διότι είναι αρκετά σαφές ως έχει. Σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση, συμμερίζομαι την άποψη υποστήριξης τροπολογίας 56. Σε σχέση με το ρόλο του Τατζικιστάν, νομίζω ότι η τροπολογία υπαριθμών 5 μπορεί να γίνει αποδεκτή, διότι θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός περιφερειακός φορέας και δράστης. Ως προς την τροπολογία 38α μετά από την παρέμβαση Επιτροπής θεωρώ ότι δεν είναι αναγκαίο να τύχει υποστήριξη, άρα θα προτείνω αύριο να μην εγκριθεί αυτή η τροπολογία. Εάν κάποιος θα ήθελε διευκρινήσεις ή άλλα τμήματα της έκθεσης, έχουμε χρόνο μέχρι την Ολομέλεια. Ωραία, με αυτή την παρέμβαση νομίζω ότι εκφράστηκαν όλα τα επιμέρους ζητήματα και έληξε και η ημερήσια διάταξη. Άρα μπορούμε να τελειώσουμε τώρα με τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. Θα βρεθούμε αύριο στις 9 εδώ σε αυτή την αίθουσα. Καλό σας βράδυ.